Αγαπητοί συνάδελφοι, λέω να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. limits, I Γιατί ήδη περιμέναμε αρκετά. Μην καθυστερήσουμε κι άλλο και δεν προλάβουμε να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμά μας που είναι κατάμεστο. Ε, καλωσορίζω όσους ε, είναι παρόντες. Ας εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Προτάσεις αλλαγής δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής. Οπότε αν δεν έχετε σχόλια, λέω να θεωρήσουμε την ημερήσια διάταξη ως εγκεκριμένη. Προχωράω στο δεύτερο σημείο, τις ανακοινώσεις της Προέδρου. Μην ξεχνάτε ότι το απόγευμα μετακομίζουμε σε άλλη αίθουσα. Θα το πω και στο τέλος βέβαια τις συνεδρία σας, το υπενθυμίσω, αλλά καλό να το έχετε υπόψη από τώρα. Και όσοι θυμάστε την πρωτοβουλία ε, έρασμος για τους τοπικούς και περιφερειακούς ερετούς, προχωράει η πρωτοβουλία αυτή. Θα σας μοιραστεί διεξοδικό σημείωμα εν ευθέτω χρόνο βρίσκεται υπό ετοιμασία. Πάντως, τα τρία θεσμικά όργανα, Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Επιτροπή των Περιφερειών, προέβησαν σε ανταλλαγή απόψεων τους τελευταίους μήνες και αποφάσισαν να κρατήσουν το φετινό προϋπολογισμό. Ούτως ή άλλως, ε, για το 2010 και 2011 είχε προγραμματιστεί ως πιλωτικό πρόγραμμα αυτό, αλλά δεν ξεκίνησε να το εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα φαίνεται ότι τα πράγματα προχωράνε κάπως και η πρόταση που συμφωνήσαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να έχουμε μια εξάμεινη δράση καταμερισμένη σε διάφορα στάδια Βρισκόμαστε τώρα σε φάση επιλογής των υποψηφίων για τη δράση αυτή και έχει ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής και μάλιστα είναι ανοιχτή για όλους τους τοπικούς ε, και περιφερειακούς ε, εκπροσώπους, ερετούς. Θα ληφθεί υπόψη και η ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων και η γεωγραφική ισορροπία οι υποψήφοι που θα επιλεγούν θα συμμετέχουν και σε μία ειδική εκδήλωση στις Open Days και θα έχουμε και επισκέψεις σε διάφορες ευρωπαϊκές περιφέρειες και πόλεις στα πλαίσια της συγκέντρωσης γνώσεων και πληροφοριών και εμπειρίες και θα έχουμε και στο τέλος ως επιστέγασμα ένα σεμινάριο. Αυτά με βάση το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπω σα είπα, έγινε συζήτηση μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων Επιτροπή Περιφερειών, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προχωράμε στην εφαρμογή του προγράμματο. Τώρα, σημείο 3, <clears throat> έκθεση Αλέν Καντέκ ίδιες πρωτοβουλίες για την στρατηγική για την περιοχή του Ατλαντικού στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον Αλέν Καντέκ, για να μας υποβάλει το σχέδιό του. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, διαπιστώνω καταρχήν με κάποια θλίψη ότι η στρατηγική για την περιοχή του Ατλαντικού δεν συναρπάζει τα μέλη της Επιτροπής μας. Πάντως ε, συναρπάζει τουλάχιστον την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Επιτροπή Περιφερειών και της ΕΡΠΕ. Ελπίζω και σε επόμενες εβδομάδες να κινήσει το ενδιαφέρον και των συναδέλφων. Πάντως ευχαριστώ τους παρόντες, γιατί υπάρχουν έστω και λίγοι παρόντες. Βέβαια, η 8η Μαΐου είναι αργία στη Γαλλία. Ίσως γι' αυτό θεώρησαν οι συνάδελφοι ότι θα πουσιάζω κι εγώ και δεν ήρθαν ούτε εκείνοι. Εν πάση περιπτώσει, κυρία Πρόεδρε, η Επιτροπή, η Επιτροπή, Περιφερειακής Ανάπτυξης μου ανέθεσε την έκθεση πρωτοβουλίας για τη στρατηγική της περιοχής του Ατλαντικού. Άλλωστε, εμείς πρωτοστατήσαμε στο σχετικό ψήφισμα του Μαρτίου του 2011 που ζητούσε μια μακροπεριφερειακή στρατηγική για την περιοχή του Ατλαντικού. Εδώ και ένα χρόνο πολλές πρωτοβουλίες έχουν αναλυφθεί και μετά από πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη ε, δεσμεύθηκαν για μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή στρατηγική ως προς τον Ατλαντικό. Και μάλιστα χαίρομαι και για την ε, ενεργό ε, συμμετοχή και κινητοποίηση των περιφερειών και των ερετών τους υπέρ αυτής της πρωτοβουλίας. Μάλιστα, θετήσαμε και μια προκαταρκτική δράση για την στρατηγική αυτή. Δημιουργήθηκε και ένα φόρουμ του Ατλαντικού και μάλιστα εκεί εκπροσωπώ εγώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το φόρουμ αυτό θα ε, ηγηθεί των προπαρασκευαστικών εργασιών και θα καταρτήσει για ένα σχέδιο δράση μέχρι τα τέλη του 2012. Αυτό το σχέδιο δράση θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με το επόμενο φυσικά πολιτες δημοσιονομικό πλαίσιο και με τις συμβάσεις εταιρική σχέση και τα επιχειρησιακά προγράμματα της πολιτικής συνοχής. Στόχος της έκθεσής μου είναι να υποβάλω προτάσεις για να εντοπίσω τις πολιτικές προτεραιότητες του σχεδίου δράσης. Ο Ατλαντικός, η περιοχή του Ατλαντικού έχει διάφορα χαρακτηριστικά. Πρόκειται για ένα δυναμικό θαλάσσιο χώρο λόγω των ανανεώσιμων θαλάσσιων πηγών ενέργεια, των θαλάσσιων μεταφορών, των αυτιλιακών κλάδων, του τουρισμού και τη αλία, καθώ και τη υδατοκαλλιέργεια. Πρόκειται για χώρο με ευαίσθητο θαλάσσιο περιβάλλον, το οποίο είναι ανάγκη να προστατευτεί. Πρόκειται για ένα χώρο που αποτελεί τη δυτική θύρα εισόδου τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το λόγο αυτό κατέχει στρατηγική θέση στην Ευρώπη. Και τέλος πρόκειται για περιφερειακό χώρο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που θέτει το ζήτημα του αμπεκλωβισμού του και της σύνδεσής του με την υπόλοιπη Ευρώπη. Τα θέματα αυτά υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα και απαιτούν την εξερεύνηση πολιτικών λύσεων στο επίπεδο των ακτών του Ατλαντικού. Θα ήθελα η στρατηγική για την περιοχή του Ατλαντικού να λάβει τη μορφή μακροπεριφερειακή συνεργασία, ώστε να ενθαρρυνθούν οι συνέργειε μεταξύ των διαφόρων μέτρων και των διαφόρων επιπέδων που παρεμβαίνουν στι πολιτικέ χωροταξικού σχεδιασμού. Η μακροπεριφερειακή λογική περιέχει επίση τη δυνατότητα συμμετοχή όλων των αρμοδίων φορέων ε, στον καθορισμό και την εφαρμογή των στόχων τη στρατηγική. Η έκθεση ζητά τη διάρθρωση τη στρατηγική γύρω από δύο θεματικού τομεί. Τον θαλάσσιο και χερσαίο χωροταξικό σχεδιασμό και την αξιοποίηση τη διασύνδεση ξηρά θάλασσα, την τόνωση του οικονομικού ιστού των περιοχών του Ατλαντικού μέσω μια βιομηχανική πολιτική προσαρμοσμένη στι ιδιαίτεροτητέ του ως προς το πρώτο θέμα, προτείνω η στρατηγική να θαρρύνει τη ε, βιώσιμη εκμετάλλευση του Ατλαντικού μέσω συντονισμένη διαχείριση όλων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που έχουν αντίκτυπο στο θαλάσσιο χώρο. Γι' αυτό προτείνω την ε, δημιουργία μιας ε, δομής προκειμένου να γίνει ένα συντονισμό με βάση διακλαδική και διασυνοριακή λογική. Θα χρειαστούμε ισχυρή δράση προκειμένου να διαφυλαχθεί η οικολογική ισορροπία και η βιοεπικιλότητα και για να περιοριστεί το αποτύπωμα άνθρακα. Στόχο τη στρατηγική θα πρέπει να είναι επίση η βελτίωση των ικανοτήτων πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων στον Ατλαντικό, ιδίω σε περιπτώσει ατυχημάτων, φυσικών καταστροφών και εγκληματικών ενεργειών. Αυτέ οι διάφορε πτυχέ θα πρέπει να ενισχυθούν με κάποια μέτρα εδαφική συνοχή. Δυστυχώ ε, αυτή η πτυχή δεν τονίζεται αρκετά στην ε, ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή του περασμένου Νοεμβρίου. Θα ήθελα η στρατηγική αυτή να συμβάλλει στον απεκλωβισμό και στην προσπελασιμότητα αυτών των περιοχών του Ατλαντικού που είναι ξόχω απόκεντρε, ειδικά μετά τη διαβρύση. Θα πρέπει να επενδύσουμε στη διασύνδεση των διαφόρων ε, δικτύων και να επενδύσουμε στην ε, ενίσχυση διασύνδεσης ε, ξηράς θάλασσας. Επίσης θέλουμε κάποιους διαδρόμους θάλασσας και υποδομές μεταφορών για να συνδεθούν οι περιοχές του Ατλαντικού με την υπόλοιπη Ευρώπη. Έρχομαι τώρα στην δεύτερη θεματική, μια βιομηχανική πολιτική για τον Ατλαντικό. Η στρατηγική θα πρέπει να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία θέσεων απασχόληση στο θαλάσσιο κλάδο. Έχουμε ένα τεράστιο οικονομικό δυναμικό εδώ σε ό,τι αφορά την γαλάζια ανάπτυξη, χάρη στις ενέργειες τη θαλάσση, την ναυπηγία, την αυτιλία, την υδατοκαλλιέργεια, τη θάλασσα. Οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να συμπληρωθούν από τις κρατικές δράσεις σε διάφορους τομείς έρευνας ανάπτυξης και ανατομίας, επαγγελματικής κατάρτισης, ανάπτυξη θυλάκων αριστείας και επενδύσεων των ΜΜΕ. Η οικονομία της θάλασσας ε, είναι κλειδί της ε, βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας. Δεν θα πρέπει να χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, διαχείριση, διακυβέρνηση της στρατηγικής. Η στρατηγική θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2014 και θα συντοριστεί με το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα αφορά όλες τις περιφέρειες του Ατλαντικού καθώς και την περιοχή της Μάχης και ε, της Ελλανδίας. Φυσικά και τις ε, εξόχως απόκεντρε περιοχές καθώς και τα διαμερίσματα, τα υπερπόντια και τις χώρες χάρη στη διεθνή συνεργασία. Θα πρέπει να συνδέσουμε τους διάφορους, να, να, να φέρουμε σε επαφή τους διαφόρους εταίρους, τις κεντρικέ τις κεντρικές αρχές, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Φυσικά έχουμε ήδη κάποια σχέδια στην περιοχή του Ατλαντικού, γίνεται ένας απολογισμός, έχουμε πολύ καλά παραδείγματα των πρακτικών, καλό θα ήταν να διδαχθούμε από αυτά. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε όλες αυτές τις εμπειρίες που έχουμε μέχρι τώρα. Τα διαρθρωτικά ταμεία και η ε, ολοκληρωμένη τέτοια πολιτική θα αποτελέσουν το τον πυρήνα αυτή τη δράση. Θα πρέπει να τη συνδυάσουμε με τι άλλε πολιτικέ έρευνε, έρευνα, ενέργεια, περιβάλλον, αλληλεία, διεθνή ε, συνεργασία, ΕΤΕ και με τι πολιτικέ των κρατών μελών καθώ και τι περιφερειακέ και τοπικέ πολιτικέ. Θα πρέπει επίση να αξιοποιήσουμε καλύτερα τα υπάρχοντα κοινοτικά κονδύλια χωρί να δημιουργήσουμε νέα δημοσιονομικά μέσα θα πρέπει να τροποποιήσουμε καλύτερα, να ε, προσανατολίσουμε καλύτερα τις υπάρξεις πολιτικές και να λάβουμε υπόψη και την περιοχή του Ατλαντικού. Επίσης, ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ε, συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα επιχειρησιακά προγράμματα και να έχουμε δική προσημείωση για τις περιοχές του Ατλαντικού. Θα υποβάλω μάλιστα σχετικές τροπολογίες στο νέο κανονισμό και τα διορθωτικά ταμεία. Επίσης, σημαντικό είναι να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα διαχείρισης του σχεδίου δράσης για να έχουμε μια νέα θηρίδα για τους δικαιούχους προκειμένου να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ των διαφόρων αρμόδιων αρχών της για τη διαχείριση των ε, ταμείων. Η στρατηγική αυτή για το Ατλαντικό αποτελεί σήμερα αντικείμενο πολιτικής συνένεση μεταξύ των κρατών μελών και των κοινοτικών θεσμικών οργάνων καθώς και των περιφερειών. Η κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συμβάλλει στο να δοθεί πνοή σε αυτό το σχέδιο Φυσικά ε, είμαι βέβαιος για την ανανέωση της εμπιστοσύνης μας και προσβλέπω σε μια ευρή υποστήριξη της έκθεσής μου. Φυσικά είμαι στη διάθεσή σας και στη διάθεση των σχεδόν εισηγητών για να συνεργαστούμε για τα σημεία που σας ενδιαφέρουν περισσότερο από την έκθεση. Ευχαριστώ, αλλά... Ας ακούσουμε τους σκιώδης εισηγητές. Κυρία Πέρας, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου καταρχάς να σας συγχαρώ κύριε Καντέκ για την εξαιρετική έκθεσή σας. Και επίσης θα ήθελα να σας ευχηθώ ε, ότι καλή επιτυχία και να σας πω ότι θα πρέπει να βασιστείτε σε μένα για αυτή την ε, πρωτοβουλία που είναι πολύ σημαντική για την περιφερειακή πολιτική. Επιτρέψτε μου τώρα να κάνω κάποιες προτάσεις, διότι θεωρώ ότι η δημιουργία μιας μακροστρατηγικής ε, ε μικροπεριφερειακή στρατηγικής για τον Ατλαντικό είναι μια καλή ευκαιρία για να αντιμετωπίσουμε τις κοινέ προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι περιοχές και οι χώρες του Ατλαντικού οι θαλάσσιες έρευνες, ε, οι λιμενικές υπηρεσίε και οι οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις. Θα ήθελα να σταθώ εν συντομία σε κάποια θέματα. Επιτρέψτε μου καταρχάς ε, να σας πω ότι πρωτίστως λείπει μια αναφορά στη σημασία του να καταφέρουμε η στρατηγική αυτή να βασίζεται σε μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση που θα υποστηρίζεται από πιο στενή συνεργασία των δημοσίων, περιφερειακών και τοπικών αρχών, των ενδιαφερομένων του ιδιωτικού τομέα και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων και των οργανώσεων και δικτύων που ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό. Γι' αυτό θεωρώ ότι το Φόρουμ του Ατλαντικού θα πρέπει να παραμείνει τουλάχιστον μέχρι το 2014 και να ενσωματωθεί ε, και να ενσωματώσει, συγγνώμη, με πιο μόνιμο τρόπο κάποιες από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές αλλά και κάποιους άλλους φορείς που αυτή τη στιγμή δεν συμμετέχουν ε, στο φόρουμ. Επίσης θεωρώ ότι είναι σημαντικό να έχουμε μια ισορροπημένη αύξηση μεταξύ των ε, εδαφών τόσο των, αλλά και των θαλασσιών χώρων και να αυξήσουμε την αστική διάσταση της μακροπεριοχής. Επίσης θα πρέπει να έχουμε και μια στρατηγική προκειμένου να θεμελιωθεί η έρευνα και η ανάπτυξη και η συνεργασία μεταξύ των ε, ερευνητικών κέντρων που βρίσκονται σε περιοχές του Ατλαντικού, ιδίως ε, σε θέματα εξειδίκευσης ε, στο θαλάσσιο και ναυτιλιακό τομέα. Τέταρτον, Όσον αφορά το θέμα της ενέργειας, θα πρέπει να υποστηρίξουμε τη συνεργασία μεταξύ των περιοχών του Ατλαντικού ώστε να θεμελιωθούν ε, πηγές ενέργειας, όπως για παράδειγμα η ε, θαλάσσια αιωλική ενέργεια ε, σε πλωτές περιοχές και την ενέργεια που έχουμε από τις θαλάσσιες περιοχές και από την, και την παλήρια. Θα πρέπει να υπάρχουν συνέργειες μεταξύ των λιμενικών ε, ε, δραστηριοτήτων, των ε, δραστηριοτήτων επιμελητίας και όλων των δραστηριοτήτων που μπορούν να ευνοήσουν τον ναυτιλιακό τομέα και θα πρέπει να υπάρχουν και δίκτυα ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και σε βιομηχανικό αλλά και σε άλλα επίπεδα στον Ατλαντικό. Επιπλέον θα πρέπει να εμείνουμε στη σημασία του να υπάρχει ένας βιώσιμος και διαρκής τουρισμός και να προστατεύεται το οικοσύστημα και η βιοποικιλότητα της περιοχής. Τέλος, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και κάποιες άλλες δράσεις ε, στον πίνακα που έχει ετοιμάσει ο συγητής, για παράδειγμα βέλτιστες πρακτικές οι οποίες μπορούν να ληφθούν υπέψη ε, κατά την ε, προετοιμασία του προγράμματος δράσης και να υπάρχει ε, κοινωνική συνοχή, το ΣΟΥΤ για παράδειγμα, ή την πρωτοβουλία για το περιβάλλον. Ευχαριστώ και συγχαίρω τον ε, κύριο Καντέκ ε, για την πολύ καλή του εργασία και να πω ότι εξ ονόματος της ομάδας μου θα παρουσιάσω κάποιες τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε Μαρία. Και τώρα... Ο Πατ Κάλαγκερ δεν είναι εδώ. Ο Φρανσουέλ Φονσί έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε οι ομάδες μας φυσικά υποστηρίζει την πρόταση. Ο Ατλαντικός ε, χώρος βεβαίω είναι ένα πεδίο στο οποίο μπορούμε να ανοίξουμε νέο περιθώριο για περιφερειακές και ευρωπαϊκές συνεργασίες. Ένα πεδίο ενδιαφέρον για μας, Γιατί όμως τον Ατλαντικό, στις περιφέρειες ε, που βρέχονται από τον Ατλαντικό, οι οποίες ε, χαρακτηρίζονται από έναν τροπισμό προς την ε, ε, πρωτεύουσα, τουλάχιστον στη Γαλλία, όλες στρέφονται προς το Παρίσι, φαντάζομαι το ίδιο συμβεί και στις άλλες χώρες. Πρέπει λοιπόν να ξεφύγουν από αυτόν τον τροπισμό οι ε, ηγετικέ προσωπικότητες των περιφερειών αυτών και να τις καθοδηγήσουν προς μια πιο αυτόνομη λειτουργία. Έτσι λοιπόν θα θέλαμε να έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση ώστε να ξεφύγουμε από τον τροπισμό αυτόν, ιδιαίτερα για τις περιφέρειες του Ατλαντικού και θα προτείνω να υπογραμμιστεί αυτό το σημείο. Ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο ε, είναι ότι οι αυτοκινητόδρομοι της θάλασσας βεβαίως είναι ενδιαφέρουσα πρόταση ωστόσο δίνουν μια εικόνα μάλλον χερσαίας μεταφοράς και δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε την, ε, το καμποτάζ, ε, την ε, μεταφορά δηλαδή την θαλάσσια μικρών αποστάσεων των εμπορευμάτων κατά τρόπο βιώσιμο με μικρές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και συμφέροντα για την οικονομία όλη αυτή η μακροοικονομική στρατηγική, ακόμη και όταν ε, αφορά διαφορετικής φύσεως θαλάσσιες λεκάνες, όπως φερειπίν τον Ατλαντικό που είναι ανοιχτή θάλασσα, σε αντιπάθεση με τη Βαλτική που είναι κλειστή, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν διαφορετικό τρόπο μακροοικονομική στρατηγική λοιπόν περιφερειακή που θα πρέπει να μας επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο καθένας να μπορεί να τοποθετηθεί σωστά στο φυσικό περιβάλλον στο οποίο διαβιώνει. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό και βέβαια υποστηρίζω την πρόταση. Ευχαριστώ κυρία Χιούπνερ. Κύριο Σταμάρση δεν είναι εδώ. Μαρή Τερέ Σμιτ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Και ευχαριστώ βεβαίως τον συναδελφό Άλαν Καντέκ, εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει και η γενικότερη δυναμική που εμφυσά στον χώρο του Ατλαντικού και υποστηρίζει διάφορα σχέδια με τον τρόπο του αυτών. Θα ήθελα να υποστηρίξω διάφορες θεματολογίες εργασία, όπως ε, η χωροταξία των θαλάσσιων και χερσαίων χωρών, χώρων καλύτερα ε, και περιοχών καλύτερη υποστήριξη και ενθάρρυνση της ε, δραστηριότητας της ζώνας της προχώμενης από τον Ατλαντικό, την εισαγωγή μονίμων ζωνών συνεργασίας και νομίζω ότι μπορεί αυτή η δουλειά να αποτελέσει πηγή έμπνευση για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε και να επιτρέψουμε την πλήρη ανάπτυξη και καρποφορία των προσπαθειών και των μέσων που διαθέτουμε. Στρατηγικές λοιπόν οι οποίες θα πρέπει να στοχεύουν στην, στην ε, χωροταξία να ενθαρρύνουν τον, ε, ε, τις επενδύσεις και τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών φορέων. Μια αντίστοιχη στρατηγική για την ε, Μεσόγειο θα πρέπει να ακολουθήσει, πιστεύω, την προσέγγιση αυτή, με ενθάρρυνση ιδιαίτερα του οικονομικού ιστού και περισσότερες δραστηριότητες. Ιδιαίτερα ο χαρακτηρισμός ε, των ζωνών στις διαπεριφερειακές αυτές δραστηριότητες που προτείνει η έκθεση θα πρέπει να ε, συζητηθεί περισσότερο. Δεν μπορούμε δηλαδή να εμποδίσουμε τη στρατηγική στις επενδύσεις ΦΕΝΤΕΡ. Ο δε στόχος για την εδαφική συνεργασία θα πρέπει να ενσωματωθεί στην, ε, στις μακροπεριφέρειες έτσι ώστε αυτές να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες και το συντονισμό που έχει εξασφαλιστεί στο πλαίσιο του στόχου 3. Ευχαριστώ πολύ. Λάσεκ. Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε και κύριοι. Θα ήθελα να πω ότι έχουμε εδώ μία πρόταση η οποία παρουσιάζει πιθανούς χώρους συνεργασίας, υποστηρίζει ξεκάθαρα συνεργατικές σχέσεις μεταξύ διαφόρων επιπέδων διαχείρισης, αλλά και μέσων νομοθετημάτων που έχουμε στη θέσή μας και Υπογραμμίζω ότι ο εισηγητή είπε τρία διαφορετικά όχι, ούτε νέα μέσα, ούτε νέα νομοθεσία, ούτε νέο προπολογισμό ζητάει. Ιδιαίτερα λοιπόν θα θέλω να υπογραμμίσω ότι μιλάει για ένα νέο πρόγραμμα δράση, πρόγραμμα δράσης το οποίο θα συμπεριλάβει τόσο το δημόσιο και το ιδιωτικό τομέα στου κόλπου του, πράγμα το οποίο θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό. Θα περιλαμβάνει φαντάζομαι δραστηριότητε από τη βάση προ τα Άρνο, που είναι και η πιο σημαντική διάσταση και ιδιαίτερα θα ήθελα να υπογραμμίσω το γεγονός ότι μια από τις, ε, ένας από τους χώρους ο οποίο αναφέρει ο εισηγητής ότι θέλει να βελτιώσει την, ε, το συντονισμό και την πρόληψη φυσικών καταστροφών και κινδύνων ε, είναι αυτό η ενίσχυση των σχετικών μονάδων. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω το εξή Πώς μπορεί ε, να γίνει η ενσωμάτωση των περιφερειακών και των άκρως απομακρυσμένων περιοχών στον στόχο αυτών. Ευχαριστώ πολύ. Όλμπριχτ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να συγχαρώ θερμότατα τον κύριο Καντέκ για το σχέδιο εκθεσής του και το συγχαίρω θερμά και εγκάρδια όχι από αυρότητα, αλλά γιατί πραγματικά το έγγραφό του είναι πολύ ισορροπημένο. Το έγγραφο αυτό αφενός υπογραμμίζει και ορίζει τους βασικούς στόχους υλοποίηση και αφετέρου προτείνει και κάποιους τρόπους δράσης. Ήμασταν και είμαστε μάρτυρες πολλών συζητήσεων για τη λεγόμενη μακροπεριφερειακή στρατηγική και γνωρίζουμε τις προσδοκίες που εγείρει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, στην έκθεση αυτή έχουμε συγκεκριμένο απολογισμό των διαφόρων στοιχείων και στην παραγράφο 22 προτείνεται τρόπος για την ε, απόκτηση αυτής της συνέργειας και προτείνει συγκεκριμένο συντονισμό των, των κοινωτικών πολιτικών στα πλαίσια του σχεδίου δράσης. Αυτό ε, δείχνει να την ανάγκη του συντονισμού. Κάτι που βλέπουμε παρακάτω ε, είναι μια αιρεσιμότητα ε, σε σχέση με την υποχρέωση ε, εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων που συνδέονται με τη μακροπεριφερειακή στρατηγική. Αυτή η κατεύθυνση που προτείνει ο συγκεκριτή είναι πολύ θετική και αποφελής. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολύ σοβαρά τη μακροπεριφερειακή στρατηγική, να ορίσουμε ρητά τους στόχους και να συνδυάσουμε τα, τους διάφορους μηχανισμούς που έχουμε στα πλαίσια της ε, Περιφερειακή πολιτική, προκειμένου με τα επιχειρησιακά προγράμματα να υλοποιήσουμε του στόχου τη μακροπεριφερειακή στρατηγική. Είναι πολύ ε, ρητή και συγκεκριμένη αυτή η κατεύθυνση και μάλιστα δεν χρειάζονται και νέα δημοσιονομικά μέσα όπως είπε και ο κύριος Βλάσεχ. Πολύ ενδιαφέρον το έγγραφο και από πολιτική άποψη πολύ ισορροπημένο. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Άννα Μιράντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς ε, να συγχαρώ τον εισηγητή για την εξαιρετική αυτή έκθεση. Και ιδιαίτερα θα ήθελα να τον συγχαρώ για το μεγάλο ενδιαφέρον, της στράτευση και την ε, έμφαση που δίνει στις ε, περιφέρειες που βρέχονται από τον Αθλαντικό. Θα ήθελα ιδιαίτερο λοιπόν να αναφερθώ στην αέναη αυτή σχέση μεταξύ κέντρου και περιφέρειας όταν προβαίνουμε σε μία προσέγγιση μακροπεριφερειακή όπως την προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει αναγκαστικά να επανεξετάσουμε τη σχέση μεταξύ κέντρου και περιφέρειας. Στην περιφέρεια του Ατλαντικού Έχουμε πρόβλημα προσβασιμότητας, πρόβλημα αναγνωρισιμότητας, αλλά και πρόβλημα συνδεσιμότητας, το οποίο ιδιαίτερο πρόβλημα συνδεσιμότητας και κοινωνικο-οικονομικής και εδαφικής συνοχής είναι αυτό που με απασχολεί ιδιαίτερο. Πρόκειται για μια έκθεση λοιπόν η οποία πιστεύω θα συμβάλλει ιδιαίτερο σε μια πιο ε, ενδιαφέρουσα, σε μια πιο ε, αποτελεσματική προσέγγιση ο κύριος Καντέκ λοιπόν προτείνει μια νέα προσέγγιση, μια νέα σωστή προσέγγιση μαζί με το πρόγραμμα πλαίσιο των διευθυντικών ταμείων, αλλά ταυτόχρονα και όλες οι αναφορές στην οικονομική συνοχή και ιδιαίτερα για τα ε, για τις περιοχές εκείνες ε, οι οποίες πλήττονται από την θαλάσσια κρίση, κυρίως από την οικονομική κρίση, αλλά κυρίως στον χώρο της θάλασσας, ε, είτε πρόκειται για ναυπηγή, είτε πρόκειται για εκτατική ή εντατική αλληλεία κτλ. Και θα πρέπει εδώ να κάνουμε διαφοροποίηση μεταξύ εκτατικής και εντατικής. Μας επιτρέπει λοιπόν να έχουμε μια πιο σημαντική πολιτική προσέγγιση και γι' αυτό και οι τροπολογίες του κυρίου Αλφόνση που θα ε, μας εμπνεύσουν και εμάς ε, θα μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε προς την συνεργασία και την διαχείριση στο περιφερειακό πλαίσιο. Θα ήθελα ιδιαίτερα ωστόσο να υπογραμμίσω κλείνοντας τους χαιρετισμούς του κυρίου Λουίς Μιγγέλ Παρίθα, εισηγητή από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος δεν μπόρεσε να έρθει, αλλά με ε, επιφόρτησε να μεταφέρω τους χαιρετισμού του, καθώς εχθές είχαμε τον κύριο Κίνγκ, τον κύριο Κουέρβο που είναι εδώ καθισμένοι, αλλά και άλλους και την υποφαινομένη ως συμμετέχουσα μόνο στη συζήτηση, μια συνάντηση για τα ίδια αυτά θέματα. Ξεσενθαρρύνω να μελετήσετε την έκθεση του κυρίου Παρίθα για την στρατηγική που πιστεύω θα συμβάλλει ιδιαίτερα στην, ε, σε μια κοινή προσέγγιση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω σου ειδικά, δεδομένου ότι υπάρχει διερμηνία θεωρώ και εγώ ότι είναι μια πολύ καλή έκθεση και ε, εντάσσεται πολύ καλά στο γενικότερο πλαίσιο των σκέψεων της Επιτροπής μας και τους βασικότερους κανόνες που θα θέλαμε να έχουμε για την περιφερειακή μας πολιτική από το 2014 και τούδε. Έχω μια ερώτηση όμως προς τον εισηγητή. Ο εισηγητής λέει ότι οι περιφέρειες γίνονται όλο και περισσότερο ενταγμένες στη διαδικασία. Γνωρίζω από τη στρατηγική της Βαλτικής ότι η μακροπεριφερειακή στρατηγική μπορεί να επιτύχει μόνο εάν η περιφέρεια ε, νιώσει ότι της ανήκει Πώς λοιπόν βλέπετε εσείς αυτό το αυξημένο ενδιαφέρον από πλευράς περιφερειών αναφέρεστε σε όλες τις περιφέρειες, διαπιστώσατε ότι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον από όλους. Ιδάλλως πώς μπορούμε να πείσουμε ε, τις περιφέρειες ε, να οικειοποιηθούν αυτή τη στρατηγική. Ευχαριστώ, δεν έχω κάποιον άλλο στον κατάλογο. Επομένως, αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να λάβει το λόγο, θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν ε, επιθυμεί να σχολιάσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι διαβάσαμε μεγάλο ενδιαφέρον την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εντάσσεται πολύ καλά ε, στο πλαίσιο των όσων προσπαθούμε και εμείς να επιτύχουμε. Η στρατηγική για τον Ατλαντικό αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας ε, στις παράκτιες περιοχές ε, και να έχουμε ανάπτυξη, ιδίως στην περιοχή του Ατλαντικού. Αποτελεί τμήμα της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντάσσεται και στην ατζέντα της Ευρώπης 2020 προκειμένου να έχουμε μια μπλε οικονομία όπως την αποκαλούμε, δηλαδή μια βιώσιμη ε, θαλάσσια και ναυτιλιακή πολιτική. θεωρούμε ότι έχει συνεισφέρει ιδιαίτερα ο κύριος Καντέκ ε, και η Επιτροπή σας ε, στο θέμα αυτό ε, σε σχέση με τα όσα ε, αναφέραμε εμεί ε, στην ανακοίνωση για την πολιτική για τον Ατλαντικό. Επικεντρωθήκαμε κυρίω ε, στα θέματα τη θαλάσσιας πολιτική και το θέμα τη ε, σύνδεσης έγινε πιο σημαντικό μετά από τις παρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των ενδιαφερομένων. Βεβαίω δεν μπορούμε να έχουμε μία καλά λειτουργούσα θαλάσσια οικονομία εάν δεν υπάρχει κατάλληλη δικτύωση και πρόσβαση στις αγορές και αυτό θα το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Επιπλέον, εξετάσαμε πολύ προσεκτικά πώς μπορούμε να διαρθρώσουμε το πρόγραμμα δράσης που ε, σκοπεύουμε να ετοιμάσουμε τουλάχιστον ως σχέδιο προγράμματος μέχρι το τέλος του έτου και τα όσα προτείνει η έκθεση θα ληφθούν δεόντως υπόψη πραγματικά μας ενδιαφέρουν οι ιδέες ε, και από κάτω προς τα πάνω και από τους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς και από τους ενδιαφερομένους και από τον, ε, ε, τους κλάδους, τους αρμόδιους. Θέλουμε ιδέες υπό την έννοια προγραμμάτων που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των νέων πολιετών ε, δημοσιονομικών προοπτικών. Και η καινοτομία στη στρατηγική αυτή είναι ότι δεν προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε του ενδιαφερομένους ε, να χρησιμοποιούν μόνο τα διαθέσιμα κονδύλιο ε, βάση του προγράμματος ε, εδαφικής συνεργασία, αλλά όλα τα ευρωπαϊκά κονδύλια, μία ταμεία, ταμείο συνοχής και κυρίω τα ερευνητικά κονδύλια του ορίζοντα 2020. Τα κράτη-μέλη που εντάσσονται, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, είναι ιδιαίτερα ενθουσιώδη και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν και τα σχετικά αρμόδια υπουργεία αλλά και οι τοπικές κυβερνήσεις για να καθορίσουμε τις βασικές ερευνητικές δραστηριότητες και προτεραιότητες και όπως σας είπα, οι ιδέες που θα δοθούν σε περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών μελών θα ενσωματωθούν ε, στις ε, συμπράξεις που θα έχουμε και ελπίζουμε να έχουμε στη συνέχεια χρήσιμα προγράμματα τα οποία θα μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε τα επόμενα χρόνια. Στο Φόρουμ του Ατλαντικού είπαμε ότι θα πρέπει να πάψει τις λειτουργίες του μετά το 2013. Αυτή ήταν μία από τις προϋποθέσεις ε, που θεωρεί το Συμβούλιο σημαντικές ε, για να προχωρήσει αυτή η στρατηγική, αλλά παρόλα αυτά θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μιας κάποιας μορφής εποπτεία ε, για να δίνονται και κατά κάποιο τρόπο κίνητρα για αυτή τη στρατηγική. Και αυτό είναι σημαντικό, διότι ε, θα πρέπει να μπορούμε να απαντήσουμε στο ερώτημα που θα μας τεθεί το 2020 τι ε, αποκομίσαμε από αυτή τη στρατηγική. Αν δεν υπάρχει μια κάποια μορφής παρακολούθηση και διοικητική εποπτεία θα είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζουμε τι ωφέλη και τι επιτεύγματα είχαμε πράγματι. Ε, γι' αυτό λοιπόν θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τους ενδιαφερομένους να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και ανάπτυξης επί τόπου και ευχαριστούμε ιδιαίτερα το Κοινοβούλιο διότι ε, είναι αυτό το οποίο υποκινεί όλη αυτή τη συζήτηση και ελπίζω ότι θα συνεχίσει να την υποκινεί και στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ο Αλέν Καντέκ νομίζω τώρα ότι θέλει να απαντήσει. Παρακαλώ. Merci, Madame la Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έλεγα εισαγωγικά ότι, ότι δεν είσαστε ε, πολύ άριθμοι. Αλλά βλέπω τουλάχιστον ότι είσαστε ε, ομόφωνοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ας αρχίσω λοιπόν να δίνω κάποιες ε, απαντήσεις στους αδέρφους, για τη Μαρία καταρχάς, που εξέφρασε ανησυχίες για το είναι διακυβέρνηση στα διάφορα επίπεδα. Είναι προφανές ότι η περιφέρεια, η κοινωνία των πολιτών συνδέεται στενά με τη διαδικασία αυτή. Είναι προφανές γιατί αποτελεί και τον κατάλληλο χώρο, το κατάλληλο επίπεδο για την υλοποίηση της στρατηγικής για τα φόρουμ, ναι, οι περιφερειακές αρχές ήδη είναι παρούσες μέσα από τα επιτροπές, συμμετέχουν στις πρώτες τους εργασίες ήδη. Στρατηγική έρευνα και τεχνολογία, θα το τα αγαπητοί συνάδελφοι, ότι όντως τη συμπεριλαμβάνουν στην έκθεση, είναι πολύ σημαντική, καινοτομία και ανάπτυξη είναι τα δύο στοιχεία στα οποία θα πρέπει να επιμένουμε ιδιαίτερω, όπως άλλωστε και στις θαλάσσιες ενέργειες και την επανεκφιαομηχάνηση στην οποία επιμένει η Μαρία που έχει πολύ μεγάλη σημασία για τι περιφερειέ μας. Ξέρουμε ότι στη διάρκεια των τελευταίων ε, ετών γνώρισαν περιοχές αυτές ε, για διάφορου λόγου, παγκοσμιοποίηση, ανάδυση των χωρών BRICS ιδιαίτερως εμφανίστηκε σημαντική απεκβιομηχάνηση και πρέπει να επιμένουμε για στην επανεκβιομηχάνηση κυρίως στο χώρο της των βιομηχανιών της θάλασσας. Βιώσιμη ανάπτυξη βεβαίω και ενσωματώνεται στρατηγική αυτή μέσω των προγραμμάτων δράσεως. Αυτές είναι οι πρώτες απαντήσεις που μπορώ να προσφέρω για τη Μαρία. Και φυσικά περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όποιε τροπολογίε έχει να καταθέσει. Ο σκιώδη ηγέτρια εκ μέρου των Σοσιαλιστών. Για τον Φρανσουά που είναι σκιώδη εκ μέρου των Πρασίνων, μου ε, σημειώνει τη συμφωνία του, άλλωστε το είχαμε συζητήσει και είχαμε συζητήσει, είχαμε συμφωνήσει καλύτερα στη διαπίστωση αυτού του τροπισμού προς την ε, πρωτεύουσα της περιφέρειας, γεγονός το οποίο διαπιστώνεται παντού σε όλες τις χώρες μας και πρέπει να διαρρήξουμε αυτή τη σχέση, αυτόν τον τροπισμό για να δώσουμε στις περιφέρειες την ενέργεια και τη δύναμη που τους ανήκει. Ε, για την οικονομία της θάλασσας όντω δεν πρέπει να αναπτύξουμε μόνο τους αυτοκινητοδρόμους της θάλασσα, αλλά να, να αναπτύξουμε, να υποστηρίξουμε και τι θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων που ιδιαίτερα υποστηρίζουν και τους στόχου του περιβαλλοντικούς και κυρίως τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Η Μαρία Τερέσα αναφέρθηκε σε μια σειρά θεμάτων, την ευχαριστώ ιδιαίτερω για τις προσθήκε στο κείμενό μου, υπενθυμίζει σημαντικά σημεία. Η υποχρεωτική επισήμανση είναι πολύ σημαντική, όπως υπόθηκε, συμφωνώ απολύτως. Ο κύριος Λάζακ έχει επίσης δώσει κάποιες σημαντικές προτάσεις. Και υπογραμμίζω ότι δεν στοχεύουμε στο να δαπανούμε περισσότερα, άλλωστε μάλλον λιγότερο να δαπανούμε παρά περισσότερα, αλλά καλύτερα αυτός είναι ο στόχος μας και χωρίς περιπλοκή των ε, διαδικασιών. Δεν θα εισαγάγουμε νέε διαδικασίε, γραφειοκρατία κτλ. Αντιθέτω, προσπαθούμε να έχουμε ένα πλαίσιο το οποίο θα μα επιτρέπει να εργαζόμαστε όσο δυνατόν πιο αποτελεσματικά με βάση τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μα και να υλοποιούμε λειτουργικά προγράμματα. Προγράμματα τα οποία θα μα επιτρέπουν να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα αμέσω. Επίση, ευχαριστώ τους συναδέλφους ε, και ιδιαίτερα για το θέμα του λειτουργικού προγράμματος. Για τον κύριο Όλμπριχτ ε, θα ήθελα να πω ότι βεβαίως θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση. Η Άννα επανέλαβε αυτή την ιδέα για τον τροπισμό τη σχέση δηλαδή μεταξύ κέντρο και περιφέρειας ε, που νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και αναφέρθηκε επίσης και στις ε, διασυνδέσεις αλλά και τις, τους οικονομικούς συσχετισμούς, τους οικονομικούς δεσμούς καλύτερα που είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν μεταξύ κέντρου και περιφέρειας. Ε, ο κύριος Γιέλσεν Νίλσον ε, έκανε κάποιες παρατηρήσεις υπογραμμίζοντας ότι θα ε, συμφωνήσει και εκείνο με, τις, ε, με την προτινόμενη έκθεση, θα την εγκρίνει, τον ευχαριστώ πολύ. Για τις περιφέρειες θέλω να υπογραμμίσω ότι διαπιστώνεται ενθουσιώδη συμμετοχή, άλλωστε έχουν εργαστεί πολύ στο θέμα αυτό και συμμετοχή στη στρατηγική αυτή για τον Ατλαντικό. Ιδιαίτερα πάντως Πρέπει να υπογραμμίσω ότι στόχος μας είναι να ενθαρρύνουμε εκείνες τις περιφέρειες που δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί. Αλλά πάντως ομολογώ ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική επαναδραστηριοποίηση των εμπλεκομένων περιφερειών, ιδιαίτερα, ιδιαίτερα στον χώρο του Ατλαντικού. Από την ε, Σκοτία μέχρι την Ανδαλουσία βλέπουμε ε, με ενθουσιασμό να συμμετέχουν ε, στις εργασίες, ιδιαίτερα στο επίπεδο της Επιτροπής των Περιφερειών, οι περιφέρειες αυτές και νομίζω ότι πρέπει να τι ενθαρρύνουμε να συμμετάσχουν στη στρατηγική των Ατλαντικών. Για να ολοκληρώσω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξήγησε τις θέσεις της. Εγώ προσωπικώς Πρέπει να πω ότι μερικές φορές στις εργασίες που έχω δώσει στο Κοινοβούλιο δεν είμαι ευχαριστημένος από τις τάσεις της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίως στο θέμα των αρμοδιότητων της Επιτροπής Αλίας. Αλλά εδώ πρέπει να πω ότι είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι. Εργαζόμαστε σε πολύ καλό πνεύμα συνεργασίας με τους συναδέλφους, ε, με τους κύριους από την Επιτροπή. Και είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια και τη συνεργασία. Εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ όλους για τις παρατηρήσεις. Από εδώ και μπρος αναπτύσσουμε τη γραπτή διαδικασία, γραπτή συνεργασία για να έχουμε πιο συγκεκριμένε προτάσεις και να ε, βελτιώσουμε την έκθεση, να την κάνουμε ακόμη πιο ενδιαφέρουσα, ακόμη πιο ουσιαστική. Σας ευχαριστώ. Περιμένω τις τροπολογίες σας και οποιαδήποτε ανταλλαγή απόψε. την Ευχαριστώ, αλλά πριν προσδιορίσουμε την προθεσμία ε, για τις τροπολογίες Ακούσαμε τον εκπρόσωπο της Επιτροπής Γενικής Διεύθυνσης ΜΑΡΕ, αλλά έχουμε και τον εκπρόσωπο της ε, Γενική, Γενικής Διεύθυνσης, ή τουλάχιστον αναπληρωτή διευθυν, Γενικό Διευθυντή της Επιτροπής Ρέγγι τον κύριο Ραμύρες. Θα μπορούσε και εκείνος να μας ε, μεταφέρει τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα ιδιαίτερο. Ε, επιδοκιμάζουμε την έκθεση του κυρίου Καντάκη για τη στρατηγική του Ατλαντικού και ασθενίζομαι πλήρως ε, τις απόψει των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Είναι γνωστή η σημασία της στρατηγικής ε, για την περιοχή του Ατλαντικού και θα πρέπει να δούμε τον αντίκτυπό της στον προγραμματισμό των διαφόρων διαρθρωτικών ταμείων στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020. Αυτή η στρατηγική προσέγγιση για την περιοχή του Ατλαντικού θα έχει επιπτώσεις στις ε, συμβάσεις εταιρικής σχέσης και στα ε, λειτουργικά προγράμματα ε, που θα δρομολογηθούν εκεί. Οπότε, σωστά αναγνωρίζετε ότι μια στρατηγική μακροπεριφερειακή ή για τις υδάτινε λεκάνες όπως είναι η περιοχή του Ατλαντικού καλό είναι να λαμβάνονται υπόψη τον προγραμματισμό και την κατανομή των κονδυλίων στις διάφορες περιφέρειες ή μεταξύ των διαφόρων λειτουργικών προγραμμάτων, επιχειρησιακών προγραμμάτων. Περιμένουμε και την έκβαση της συζήτησης και την τελική διαμόρφωση της έκθεσης και εμείς θα φροντίσουμε να εκπονήσουμε ένα κατάλληλο σχέδιο δράσης που να επιτρέπει την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής. Οπότε η μοναδική απόφαση που μπορούμε να λάβουμε σήμερα είναι για την προθεσμία των τροπολογιών. Προτείνω μέχρι τις 15 Μαΐου, 12 το μεσημέρι, μία εβδομάδα ακόμη δηλαδή μας απομένει. 15 Μαΐου, 12 το μεσημέρι, λίγη διορία για την υποβολή των τροπολογιών. Ολοκληρώνουμε το σημείο 3 και τώρα έχουμε μια σπάνια κατάσταση όπου έχουμε ένα κενό μισής ώρας, γιατί δεν μπορούμε να συζητήσουμε κάποια απογευματινά θέματα, λείπουν οι συνάδελφοι. Οπότε το μόνο που μας απομένει είναι να διακόψουμε για 25 λεπτά τη συνεδρίασή μας και να ξαναδώσουμε ραντεβού εδώ στις 10 και 25 προκειμένου να συνεχίσουμε τη συζήτηση με τους πρόεδρους των τριών σημαντικότερων τοπικών και περιφερειακών οργανώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία μικρή διακοπή λοιπόν και ραντεβού στην αίθουσα και πάλι σε 20 λεπτά. Dear Συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε για να ξαναρχίσουμε. Καλημέρα σας και πάλι. Ιδιαίτερα καλωσορίζω και χαιρετίζω τους προσκεκλημένους μας. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε απευθείας αναμετάδοση. Γι' αυτό μην το ξεχνάτε αυτό όταν μιλάτε. Προσπαθείτε να χαμογελάτε που και που και να δίνετε ωραία εικόνα. Έχουμε μία ε, έκτακτη κατάσταση εδώ γιατί δεν συνηθίζουμε να συνεδριάζουμε παρουσία των προέδρων των βασικότερων στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιφερειακών οργανώσεων στην Ευρώπη. Αυτά στα πλαίσια του νέου δημοσιονομικού πολίτους πλαισίου 2014-2020. Να σας υπενθυμίσω ότι ήταν πρωτοβουλία των συναδέλφων από τις περιφερειακές οργανώσεις και κυρίως του Ζαΐν Βλεντριά, του Πρόεδρου της Διάσκεψης των Απομακρυσμένων και Θαλάσσιων Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, CPMR, e ε, ήταν πολύ δραστήριος ε, για την οργάνωση αυτής της ε, συνάντησης και χαιρόμαστε που είστε εδώ για να μας κάνετε και μια παρουσίαση προσώπος. Έχουμε λάβει φυσικά τα, διάφορα, τα διάφορα έγγραφα της οργάνωσής σας, αλλά το ότι θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα απευθείας ε, συζήτησης, ε, ανταλλαγής απόψεων και διασκέδες κάποιων αφιβολιών είναι πολύ ευχάριστη. Μάλιστα, Έχουμε και μια προθεσμία μέχρι το Μάιο για να υποβάλουμε τροπολογίε. Ε, ε, και θα έχουμε και μια προκατακτική ψηφοφορία, ψηφοφορία ανατολισμού τον Ιούλιο για τον σχετικό κανονισμό. Μάλιστα, προτείνεται μέχρι τέλη του έτους ε, η υιοθέτηση του νέου κανονιστικού πλαισίου. Βέβαια, θα εξαρτηθεί αν θα διαλύσουμε το χρονοδιάγραμμα και από τις διαπραγματεύσεις ε, για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και τον προϋπολογισμό. Δεν μπορούμε εμείς να ολοκληρώσουμε το έργο μας για τους κανονισμούς αν δεν ληφθούν οριστικές αποφάσεις για τη χρηματοδότηση. Πάντως κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποφύγουμε καθυστερήσεις ε, ως προς την εφαρμογή των νέων δημοσιονομικών προοπτικών από το 2014. Οπότε θα ήθελα να καλωσορίσω τους εκπροσώπους και των τεσσάρων οργανώσεων, τον Ζω Ιβ Λεντριάν, τον πρόεδρο της διάσκεψης των απομακρυσμένων και θαλάσσιων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, κύριε Μισελ Σαμπάμ που είναι πρόεδρος συνέλευση των περιφερειών της Ευρώπης, καλώς ήρθατε. Ε, μετά εκ μέρους του, Προέδρου, του Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης θα έπρεπε να έρθει κανονικά ο πρόεδρος, ο κύριος Βόλφκαν Σούστερ, αλλά τον αντικαθιστά η κυρία Κάρλαν ε, Γκούναρσον, που είναι πρόεδρος των θεματικών πλατφορμών για η φόρο τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη του Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης. Καλώ ήρθατε κυρία Γκούναρσον και κύριος Πολ που είναι μέλος εκτελεστικής επιτροπής ε, του EuroCities. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Θα σας δώσω λοιπόν το λόγο στους ε, τέσσερις σας παρακαλώ, να μην ξεπεράσετε το 15 λεπτό στις ε, παρουσιάσεις σας, ώστε να μας μείνει λίγο ο χρόνος για υποβολή ερωτήσεων και παρουσίαση των δικών μας σχολείων και παρατηρήσεων. Θα ήθελα λοιπόν πρώτα να δώσω το λόγο στον κύριο Jean-Yves euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρία Πρόεδρε, να ξεκινήσω την ομιλία μου, γιατί πρέπει να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μας απευθύνατε, να προβούμε σε ανταλλαγή μαζί σας απόψεων για το νομοθετικό πακέτο για την πολιτική συνοχή. Η διάσκεψη των θαλάσσων περιφερειακών περιφερειών εργάζεται σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάνω στο θέμα αυτό από την δημοσίευση των νομοθετικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον προηγούμενο Οκτώβριο και με χαρά ερχόμαστε να σας προσφέρουμε επικοδομητικά επιχειρήματα πάνω στο σημαντικό αυτό θέμα τα οποία απορρέουν από την εμπειρία και τη συνεργασία τη περιφέρειας και τη τοπική μας οργανώσεις. Έτσι λοιπόν και καθώς πια έχει προχωρήσει η κατάσταση και δεν μπορούμε να περιζόμαστε μόνο σε δηλώσεις, έχουμε καταθέσει ε, ως εκπρόσωποι των ενώσεων των περιφερειών, των τοπικών αρχών της ε, Ευρώπης, προτάσεις συγκεκριμένες μετροπολογίες για να σας βοηθήσουμε στην προσπάθειά σας, στη βελτίωση της συνολικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καθώς λοιπόν όλοι διακαώς υποστηρίζουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, αποφασίσαμε και εμείς να ακολουθήσουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Εγώ προσωπικώς τώρα θα σας εκθέσω τα θέματα τα σχετικά με την υπαγωγή σε όρους. Μετά θα δώσω το λόγο στην κυρία Σαμπό για την θεματική συγκέντρωση. Μετά η κυρία Γκούναρσον θα μιλήσει για τις εταιρικές σχέσεις και την πολυεπιπεδική ε, διακυβέρνηση και μετά ο κύριο Στίλσλεϊ από το EuroCities ε, θα ολοκληρώσει την σύνοδο, τη δική μας παρέμβαση με το θέμα των αστικών κέντρων και του πακέτου της συνοχής. Πριν όμως ε, εκθέσω τις δικές μου θέσεις στο πρώτο σημείο, θα ήθελα να επισημάνω ότι σε όλες μας τις πάρεμβάσει συμφωνούμε ευρέως με την προσωρινή έκθεση της κυρίας Κρέλ και του κυρίου Φανίστηλ Ρόι που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο. Την ε, θεωρούμε λοιπόν πρόσφορη την έκθεση αυτή. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τη δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα. Ιδιαίτερος για τις προσεγγίσεις αυτές οι οποίες ε, ε, είναι σύμφωνες με τις προσδοκίες των περιοχών μας. Θα ήθελα να ξεκινήσω λοιπόν με την υπαγωγή σε όρους, μακροοικονομικούς όρους. Συμφωνούμε με τη θέση που επικρίνει το σύνδεσμο που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταξύ των επιδόσεων που σχετίζονται με την υλοποίηση, με την εφαρμογή μάλλον των, ε, ή την χρήση των διαδροτικών πόρων και τι μακροοικονομικέ τις μακροοικονομικές επιδόσεις των κρατών μελών. Ιδιαίτερα συμφωνούμε με τη διαπίστωση την οποία, στην οποία προβαίνεται και ίσως προς τον αθέμητο χαρακτήρα τιμώρηση των μέτρων υπαγωγή σε όρου, μακροοικονομικού όρου που αποβαίνουν βάρο των περιφερειών και δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί θα πρέπει αυτοί οι όροι να εφαρμόζονται μόνο στην πολιτική συνοχή και όχι στι λοιπού χωρού ή τομεί του ε, κοινοτικού προπολογισμού. Και επίσης, δεδομένων των δημοσιονομικών συνθήκων και την, που επισημάνατε και εσεί, κυρία Πρόεδρε κατά την εισαγωγή σα και της λογιστικής προσέγγισης που φαίνεται να υπαγορεύει τι διαπραγματεύσει επέδο Συμβουλίου, εμείς θα θέλαμε να προετοιμαστούμε για το ενδεχόμενο ε, μακροοικονομική όρη εν τέλει, παρότι δεν συμφωνούμε με την ιδέα αυτή, ε, εισαχθούν στο, στο νομοθετικό πλαίσιο και γι' αυτό θα θέλαμε να προτείνουμε τροπολογίες ε, επί του άρθρου 21 του Γενικού Κανονισμού για τους μακροοικονομικούς όρους, όρους μακροοικονομικών επιδόσεων και συγκεκριμένα οι προτάσεις μας ε, είναι οι εξής. Σε περίπτωση άρσης ε, των διαρθρωτικών ταμείων αυτή πρέπει να αφορά μόνο τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις και όχι τις πληρωμές, πράγμα το οποίο δεν θα επηρέαζε εν έργα και θα επέτρεπε στις αρχές διαχείρισης να αναπρογραμματίσουν ε, τα κονδύλια που έχουν στη θέση τους κατά τρόπο τακτικό, χωρίς να επηρεάζονται λοιπόν οι πληρωμές, άρα πρέπει να διαγραφεί ο όρος πληρωμές από το άρθρο 21. Δεύτερον, η Επιτροπή θα πρέπει αυτομάτως ε, να συνδέει και να, να συνδέεται και να συνεργάζεται με τις αρχές διαχείρισης των ευρωτικών ε, ταμείων για να βοηθήσει σε όποιες τροποποίησεις χρειάζονται σε, μέσα στα προγράμματα αυτά. Προτείνουμε μια τροποποίηση με εισαγωγή νέας παραγράφου στο σχετικό σημείο. Και τρίτον, προτείνουμε ένα το επίπεδο, ένα, μια οροφή δηλαδή, για το επίπεδο άρσης των δεσμεύσεων που υπολογίζονται επί του ΑΕΠ, του εν λόγω κράτου μέλου, όπω γίνεται τώρα και με το Ταμείο Συνοχή, και ω εκ τούτου οι μακροοικονομικοί ε, όροι δεν θα επηρέαζαν προγράμματα, ε, τα προγράμματα παρά μόνο κατά τρόπο αναλογικό και όχι απόλυτο. Γι' αυτό λοιπόν ε, καταθέτουμε τις προτάσεις μας, είμαστε διάθεση σας για να τις συζητήσουμε και χωρίς να θέλω να επεκταθώ υπερβολικά σε ένα έγγραφο το οποίο είναι μόνο έγγραφο εργασία προ το παρόν που μόλις δημοσιεύθηκε, θα ήθελα όπω και εσεί αγαπητοί συνάδελφοι να επισημάνω πω θεωρούμε το έγγραφο αυτό σημαντικό, θεωρούμε ότι έχει πολύ σημαντικό ρόλο να διδραματίσει για να βελτιώσει τον συντονισμό και την ολοκλήρωση των διευθυντικών ταμείων όπω και εσεί θα θέλαμε το έγγραφο αυτό, το κείμενο αυτό να προσαρτηθεί ω παράρτημα στο γενικό κανονισμό και όχι ε, να έχει τη μοίρα ενός νομοθετικού κειμένου κατεχώρηση πράξεως όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί, και ε, σας εξηγώ λοιπόν ότι θεωρούμε ότι θα πρέπει το έγγραφο αυτό να υπάγεται σε πραγματεύσεις ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως και οι προτάσεις των κανονισμών που σχεδεύονται με το πακέτο αυτό της Επιτροπής. Δεύτερον, οι ειδικοί μας σε θέματα διαχείρισης, αρχών διαχείρισης μας εξηγούν ότι μπορεί η κατεχώρηση πράξης να προξενήσουν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ε, σύγχυσης, πολύ μεγαλύτερο μάλιστα από ό,τι γνωρίζουμε τώρα, ενώ η προσπάθειά μας είναι να προστεύσουμε τις διαδικασίες. Και τρίτον και τελευταίον, για το σημείο αυτό, Πιστεύουμε ότι είναι πολύ πιο ε, συνεκτικές οι προτάσεις ε, για το στρατηγικό κοινό στρατηγικό πλαίσιο για το συντονισμό των ταμείων και τον γενικό κανονισμό για τα ερωτικά ταμεία ε, από το γενικό πλαίσιο. Επίση, ενισχύουμε ιδιαίτερω για ορισμένε από τι προτάσει ε, του Γενικού Στρατηγικού Πλαισίου, του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου, που θεσπίζουν ε, σύνδεσμο μεταξύ των διευθυντικών ταμείων και την οικονομική διακυβέρνηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Κοινό Στρατηγικό Σχέδιο δεν θα πρέπει, που δεν είναι να μετατραπεί σε εργαλείο το οποίο θα, παραβλα... θα παρέβλαπτε ενδεχομένω την ε, πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και τον πολυετή προγραμματισμό των ταμείων και τη πολιτική συνοχή. Το να επαχθεί λοιπόν ο προγραμματισμό των ταμείων στον κύκλο τη οικονομική ευρωπαϊκή διακυβέρνηση ενισχυμένο και με συγκεκριμένες συστάσεις ανακράτος μέλος θα σήμαινε ουσιαστικά την αμφισβήτηση των ίδιων των ε, θεμελίων της πολιτικής συνοχής και της νομοποίησης της μακροπρόθεσμα. Και γι' αυτό προτείνουμε ότι οι συμβάσεις εταιρική σχέση και τα προγράμματα, τα λειτουργικά προγράμματα δεν θα πρέπει πουθενή, ε, δεν θα πρέπει να εξετάζουν αποκλειστικά και μόνο τις ε, συστάσεις, ειδικές συστάσεις ανακράτους κατά την φάση ανάπτυξης, παρά μόνο στην αρχή της περίοδου προγραμματισμού, σύμφωνα με το 87 του Γενικού Κανονισμού και όχι κατά ε, ετήσια περίοδο πράγμα το οποίο θα ε, σήμαινε σεβασμό βέβαια του, της αρχής του πολιετούς προγραμματισμού. Για να ολοκληρωθεί το κεφάλαιο για, τις, ε, για τους όρους, θα ήθελα να σας ε, ενημερώσω για την πρότασή μας σε σχέση με την υπαγωγή σε όρους εξ άντε εκ των προτέρων, με ιδιαίτερη ικανοποίηση με το γεγονό ότι το Συμβούλιο και η έκθεση κυρίας Καρέλ και του κυρίου Φαναντή Ροϊ υπογραμμίζουν ότι υπογραμμίζουν ότι η αναγκαιότητα αυτή οι όροι, οι εκ των προτέρων, οι εξάντε, ε, να έχουν ε, συνέπεια, να έχουν ε, συνάφεια, άμεση συνάφεια με τα διορθωτικά ταμεία, πράγμα το οποίο είναι σύμφωνα και με τις δικές μας θέσεις και υπογραμμίζουμε ιδιαίτερως ότι θα πρέπει οι όροι εξάντε να ε, έχουν σαν κύριο μοναδικό στόχο τη βελτίωση τη αποτελεσματικότητα πολιτική συνοχή. Πολλού από του όρου προτείνονται αφορούν ότι γενικότερη προσαρμογή στην νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, πράγμα το οποίο δεν μα φαίνεται ε, σωστό και απαραίτητο και Μεγάλο αριθμό των προποθέσεων εξάντε, γενικών προποθέσεων εξάντε από το παράρτημα 4 του Γενικού Κανονισμού προτείνουμε να καταργηθεί όταν αυτές έχουν ε, να κάνουν με όταν αυτές οι προϋποθέσεις έχουν να κάνουν με την εγγύηση της μεταφοράς ε, και τη εφαρμογή των οδηγιών η περίοδος για την εφαρμογή θα πρέπει να παραταθεί ως την 31η Δεκεμβρίου του 2017 έτσι ώστε να αποφευθεί κάθε επιπλέον ε, βάρυνση γραφειοκρατική στην περίοδο προγραμματισμού και ιδιαίτερα αναφερόμαστε στην τροποποίηση του άρθρου 87 του κανονισμού. Θα ήθελα κλείνοντα. να αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο σημείο στο πεδίο εφαρμογή του ΦΕΝΤΕΡ, Ταμείο Περιφερειακή ανάπτυξη, στο άρθρο 3 συγκεκριμένου του ειδικού κανονισμού, και ιδιαίτερα καθώς υποστηρίζουμε την ιδέα, της, την αρχή της θεματικής συγκέντρωσης των εξωτικά ταμεία γενικότερα, ε, και παρότι μάλλον υποστηρίζουμε αυτή την αρχή, βλέπουμε από την εμπειρία μας ότι θα ήταν ε, σκόπιμο να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογή του ΦΕΔΕΡ για να ε, συμβάλλει στη χρηματοδότηση έργων υποδομής στις περιφέρειες και τι πιο πλούσιες και αυτό το λέω ιδιαίτερο, καθώς το ΦΕΝΤΕΡ ιδιαίτερα αυτή την εποχή έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει ως ε, μέσο μόχλευσης για να ε, προσελκύσει στις διάφορες περιφέρειες ιδιωτικές επενδύσεις και ιδιαίτερα ε, επενδύσεις στο ίντερνετ υψηλής ε, ταχύτητας και αυτός είναι ο ιδιαίτερος λόγος για τον οποίο καταθέτουμε τη συγκεκριμένη πρόταση. Δεύτερον, το ΦΕΝΤΕΡ έχει σημαντικές περιβαλλοντικές, σημαντικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο σε ορισμένε περιφέρειες, ιδιαίτερα όσον αφορά την εξασφάλιση επενδύσεων και λύσεων μεταφορών βιώσιμου χαρακτήρα στις πόλεις και τις, στα αστικά κέντρα και την περιφέρεια. Επίσης, ορισμένες περιφέρειες που αντιμετωπίσουν ιδιαίτερες δυσκολίες ή μειονεκτική θέση, όπως περιφερειπίν ε, στις σκανδιναβικές περιοχές ή τις νησιωτικές, μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν λοιπόν αυτές τις περιφέρειες στο ΦΕΝΤΕΡ για να ισοσταθμίσουν αυτές τις ιδιαίτερες ανάγκες που έχουν. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θέλουμε να καταργηθεί η παράγραφα στο άρθρο 3 του κανονισμού ΦΕΝΤΕΡ που περιορίζει το πεδίο εφαρμογή του στις πλέον ανεπτυγ... στις ε, λιγότερο ανεπτυγμένες ε, περιοχές. Θα δείτε περισσότερα παραδείγματα λοιπόν ε, όλων αυτών στο, στο δικό μας έγγραφο με τις προσκεκριμένες προτάσεις τροποποίησης για το πακέτο της συνοχής που σας έχουμε διαμενήμει και βεβαίως ε, ελπίζουμε ότι θα έχουμε την ευκαιρία να ξανασυστήσουμε τα σημεία αυτά στη συζήτηση που θα ακολουθήσει με τις παρεμβάσεις των Προέδρων των λοιπόν οργανώσεων. Δίνω το λόγο στη κυρία Σαμπάν ζητώντα και συγγνώμη για τη βραχνισμένη μου φωνή. Ευχαριστώ πολύ. Ο Μισελ Σαμπάτο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, και Ευρωβουλευτέ. θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση στη συνεδρίαση και θα ήθελα εκ μέρους της Συνέλευσης Περιφερειών της Ευρώπης να σας μεταφέρω τις απόψεις των μελών μας για το νομοθετικό πακέτο του επόμενου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Η συνέλευσή μας δίνει ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το σχέδιο και σε αυτή την πολιτική. Και μάλιστα στην Αυστρία το περασμένο ε, Δεκέμβριο ε, υποβάλαμε το μανιφέστο μας στην Πολωνική Προεδρία και στον Επίτροπο Χαν. Επιμείναμε στο γεγονός ότι η πολιτική συνοχή θα πρέπει να, να παραμείνει μια ολοκληρωμένη και ελαστική πολιτική που θα εντάσσεται σε μια συνολική εδαφική στρατηγική. Θα πρέπει να έχει ως στόχο τη βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας και τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων ε, στο εσωτερικό της κάθε περιφέρειας. Με άλλα λόγια, επειδή οι περιφέρειες, τα εδάφη είναι διαφορετικά μεταξύ τους, επειδή έχουν διαφορετικά, διαφορετικό δυναμικό και επειδή έχουν τις ιδιαιτερότητες, τις αδυναμίες και τους ιδιάζοντες στόχους τους, θα πρέπει να αναμειγνύονται και σε πρώτερο στάδιο, στον προσδιορισμό των στόχων, στην εφαρμογή των προγραμμάτων των κοινοτικών ταμείων, αλλά και σε τελικό στάδιο στη φάση αξιολόγησης των διαφορών σχεδίων και προγραμμάτων στα πλαίσια της γενικής στρατηγικής. Αυτή είναι η φιλοδοξία μας για την πολιτική συνοχή. Σημαίνει ότι είμαστε σύμβατοι με τη συγκέντρωση των ταμείων, όπως προβλέπεται στο κοινοπλαίσιο στρατηγικής ή ως προς τις ε, δράσεις ε, κλειδιά. Το αντίθετο πιστεύω, γιατί είναι σημαντικό να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητές μας, ε, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της κρίσης που διανύουμε. Είναι επίσης σημαντικό, ουσιώδου σημασία θα έλεγα, μεσούσης της κρίσης, να δούμε τι περιμένουν οι πολίτε από εμά και τι προσδοκούν από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα, γιατί αυτό που ζητούν ουσιαστικά είναι μια πιο εύρωστη και μια πιο αηφόρο ανάπτυξη. Φάνηκε αυτό του τελευταίου μήνε. Επίση, για να είναι η θεματική συγκέντρωση επιτυχημένη, θα πρέπει να δώσουμε έμφαση σε μερικέ ασφαλιστικέ δικλείδε. Σημείο πρώτο, θα πρέπει να αφήσουμε στις περιφέρειες το απαραίτητο περιθώριο λιγμών για να εφαρμόσουν πολιτικές που θα έχουν νόημα στη δική τους επικράτεια. Και τα μέτρα της θεματικής αυτής θα πρέπει να τα ανταποκρίνονται φυσικά στους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη του 2020. Δεν θα πρέπει να επαναλάβουμε τα λάθη της ε, στρατηγικής της Λισαβόνας, που ε, μετέτρεψε την ηθίκη αφόρα ανάπτυξη σε έναν ευσεβή υπόθεκη, όχι, όχι σε αποτελεσματική πολιτική. Θα πρέπει να είμαστε χρήσιμοι και σε τοπικό επίπεδο. Οπότε οι νευραλικέ δράσει θα πρέπει να είναι ενδεικτικέ και να δίνουν τροφή για σκέψη στι περιφερειακέ και τοπικέ αρχέ, προκειμένου στα πλαίσια των ε, συμβάσεων εταιρική σχέση να δουν τι ανταποκρίνεται καλύτερα στι εδαφικέ του ιδιαιτερότητε δεν θα πρέπει να επιβάλλουμε ελαστικά, ανελαστικά συγγνώμη, και ομοιόμορφα μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό δεν έχει νόημα. Το να επιβάλλουμε εκ των άνω μεταρρυθμίσει αντί να στηρίξουμε εδαφικές ε, περιφερειακές πολιτικές ε, ε, δεν έχει νόημα. Υπάρχουν πολύ σημαντικοί κίνδυνοι, καθόλου αμεληταίοι, που τους γνωρίζετε και ε, ελοχεύει ο κίνδυνο να καταλήξουμε στο αντίθετο από το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Ο πρώτο κίνδυνο είναι οι περιφέρειε να παραγωνίσουν του κανόνε, να του παραμερίσουν και παρόλα αυτά να υποστηρίξουν, να συνεχίσουν ε, τα τοπικά του προγράμματα που δεν θα έχουν όμω αναγκαστικά μια προστιθέμενη αξία. Για παράδειγμα, η οικοδόμηση κρατικών ε, δημόσιων κτηρίων χαμηλή κατανάλωση είναι ήδη προτεραιότητα στα προγράμματα δόμηση των διαφόρων περιοχών. Ποια θα είναι όμως η προστιθέμενη αξία. Ε, επίσης, δεύτερος κίνδυνος είναι τα διάφορα προγράμματα να μην ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των περιοχών, κάτι που θα οδηγήσει σε κατασ... κατασπατάληση των πόρων και η μερική αποτυχία των εξεχρονισμού των υποδομών ε, μεταφορών ε, στα, στα λιμάνια, όπως υποσήμανε η... Ε, το ελεκτικό συνέδριο, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στα άρθρα 10 και 11 του κανονισμού, του κοινού κανονισμού, προτείνουμε πριν τις δράσεις κλειδιά να προσθέσουμε το ενδεικτικές, το επίθετο ενδεικτικές. Είναι σημαντικό να έχουμε κάποιες προτεραιότητες, αλλά δεν μπορούμε να επιβάλλουμε αναλαστικά και σε όλους τα ίδια μέτρα. Δεύτερο σημείο, το θέμα της θέσης που έχουν οι διάφορες ε, περιφέρειες ε, σε ό,τι αφορά τα, τα, τα θέματα των συμβάσεων εταιρική σχέση. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε κατά τη θεματική συγκέντρωση. Το αντίθετο. Οι περισσότερε περιφέρειε ε, είναι υπέρ τη ε, ε, εστίαση σε περιορισμένο αριθμό πολιτικών προτεραιοτήτων. Και μάλιστα κάποιε περιοχέ το κάνουν ήδη. Ε, όπως όμως τα κοινοτικά θεσμικά όργανα δεν μπορούν να επιβάλλουν ομοιόμορφα μέτρα σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια, είναι επιτακτική ανάγκη τα κράτη-μέλη να μην ε, επιβάλλουν περιορισμένο αριθμό προτεραιοτήτων ε, σε εθνικό επίπεδο και μάλιστα προτεραιοτήτων που έχουν προκαθοριστεί. Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση θα πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε φάση εφαρμογής ενός προγράμματος και σχεδίου, γιατί οι περιφέρειες είναι οι κατάλληλες να αποτιμήσουν τις δυσκολίε, τι αδυναμίε, την ισχύ του και το δυναμικό ανάπτυξή του. Χωρί κάτι τέτοιο η θεματική συγκέντρωση δεν θα αποφέρει καρπού και δεν θα εξυπηρετήσει το στόχο της εξασφάλισης μεγαλύτερης εδαφικής συνοχής. Ο κίνδυνος είναι τεράστιος να καθορίσουν τα κράτη-μέλη μόνοι τις προτεραιότητες, να τις κατανέμουν βάσει τη στρατηγική τους στις διάφορες περιφέρειες, χωρίς να είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους, ούτε καν στο δυναμικό τους, κάτι που είναι πολύ χειρότερο. Επίσης, θα πρέπει να προσδιορίσουμε κάποιες ε, προτεραιότητες ε, σε περιφερειακό επίπεδο και να γίνει συγκέντρωση σε εθνικό επίπεδο. Στο τελευταίο έγγραφο εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ανάγκη ε, ανάμειξης των περιφερειών σε πρώτερο στάδιο της επεξεργασίας των προγραμμάτων επισημαίνεται. Βέβαια, είναι το πρώτο μόνο σημείο. Προτείνουμε στο άρθρο 16 του κοινού κανονισμού να διευκρινιστεί ότι τα κράτη-μέλη ε, ε, έχουν πλήρη εταιρική σχέση σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των προγραμμάτων με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές με βάση τις ανάγκες των περιφερειών. Τρίτο και τελευταίο σημείο. Η θεματική συγκέντρωση στη Στρατηγική Ευρώπη του 2020 θα πρέπει σε καμία περίπτωση να μας κάνει να μελούμε τον πρωταρχικό στόχο των ταμείων του στρατηγικού πλαισίου το κοινό στρατηγικό πλαίσιο που είναι η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή η εδαφική προοπτική θα πρέπει να περιλαμβάνεται στις κατευθυντήρες γραμμές του προγράμματος. Δηλαδή θα πρέπει να αξιοποιήσουμε το κεφάλαιο και, τις, ε, και το δυναμικό της κάθε επικράτειας, του κάθε, της κάθε περιφέρειας και να μην έχουμε μια ομοιόμορφη λύγηση για όλου. Η συνέλευσή μα ζητά το άρθρο 9 του κοινού κανονισμού να συμπληρωθεί με τον εξή τρόπο. Κάθε ταμείο που εμπίπτει στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο στηρίζει του θεματικού του ακόλουθου στόχου σύμφωνα με την αποστολή του, προκειμένου να συμβάλλει στην υλοποίηση τη στρατηγική τη Ένωση για μια ευφυή, αηφόρο ε, και ανάπτυξη χωρί αποκλεισμού και να υλοποιήσει του του στόχου συνοχή που προσδιορίζει το άρθρο 117 τη συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να συνδυάσουμε τη θεματική συγκέντρωση της στρατηγικής του 2020 με την ε, φιλοδοξία μιας καλύτερης εδαφική συνοχή στα πλαίσια της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης την πεποίθησή μας και απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της επόμενης πολιτικής συνοχής. Θα αποτελέσει ένα σημαντικό μόχλο αποτελεσματικής ανάπτυξης μόνο εφόσον συμβάλλουν σε αυτήν και οι τοπικές και περιφερειακές οργανώσεις και αρχές. Ευχαριστώ κυρία Σαμπάν. Θα ήθελα να ζητήσω από την ε, κυρία Γκούνερσον να μιλήσει εκ μέλους ε, των Ευρωπαϊκών ε, Δήμων και κοινοτήτων. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Και σας ευχαριστούμε που μας προσκαλέσατε σε αυτή τη συνεδρίαση. εκπροσωπούμε το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και είναι πολύ καλή ευκαιρία για να σας παρουσιάσουμε τα σημεία τα οποία θεωρούμε αναπόσπαστο τμήμα. Η CEMR εκπροσωπεί πάνω από ε, χίλιους δήμους και κοινότητες σε, διαφορετικές, σε 40 διαφορετικές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γεγονός που σημαίνει ότι κάνουμε μία απόπειρα να εκπροσωπήσουμε τα συμφέροντα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο όπως και οι συνάδελφοι που εκπροσωπούν τις οργανώσεις τους εδώ σήμερα. Αν δούμε την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, έχει γίνει πλήρης έρευνα και αξιολόγηση στα κράτη-μέλη και εξετάσαμε τις ε, επιδράσεις ε, των ε, εργασιών που προέκυψαν από το Διαρθρωτικό Ταμείο, εξετάσαμε τα οργανωτικά ζητήματα και την εφαρμογή και πρέπει να εξάγουμε τώρα τα συμπεράσματά μας και το τι μας αποδεικνύουν. Όπως έλεγε και ο κύριος Σαμών πριν από λίγο, η στρατηγική της Λισαβόνας δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιτυχία. Και αυτό για πολλούς λόγους. Ένας λόγος είναι διότι το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο δεν είχαν πλήρη εμπλοκή στο ζήτημα. Όταν λέω λοιπόν ότι πρέπει να εξάγουμε τα συμπεράσματά μας, νομίζω ότι ε, το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η στρατηγική της Λισαβόνας είχε ελάχιστη επιτυχία και αυτή τη στιγμή, στην τρέχουσα περίοδο, όλα τα κράτη-μέλη βιώνουν κρίση. Η νέα λοιπόν προγραμματική περίοδος επικεντρώνεται στη Στρατηγική Ευρώπη 2020, την ευφυή e e, βιώσιμη ανάπτυξη για όλους και την εδαφική ατζέντα. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα για τις μελλοντικές ε, προοπτικές για την επόμενη προγραμματική περίοδο, εάν συμμετέχουν και το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Θα ήθελα να σταθώ στην αρχή της εταιρική σχέσης. Εμείς ε, στο CMR e υποστηρίζουμε στεναρά αυτή την αρχή και θεωρούμε ότι είναι μια γενική προσέγγιση και όχι μόνο μια γενική αρχή. Είναι η γενικότερη προσέγγιση που θα πρέπει να έχουμε στην ευρωπαϊκή πολιτική και είναι και μια αρχή που επηρεάζει το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο σε πολύ σημαντικό βαθμό. Έχουμε μια πολύ θετική εικόνα της έκθεσης του κυρίου Φανίστερ Ρόι, όπου προτείνεται να γίνουν κάποιες προσθήκες ε, και εκεί διαπιστώνουμε ότι τα όσα ε, πρεσβεύουν το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο έχουν ληφθεί όντω υπόψη. Αυτό όμω, το οποίο μα ενδιαφέρει περισσότερο είναι να συμμετέχουν πλήρω οι τοπικέ και περιφερειακές αρχές, όχι μόνο κατά την προπαρασκευαστική περίοδο του προγράμματο και όχι μόνο κατά την προετοιμασία των ε, ε, συμβάσεων εταιρική σχέση. αλλά και σε όλα τα επόμενα στάδια της εφαρμογής της πολιτικής συνοχής. Εξετάζοντας το σχέδιο έκθεσης ε, των κυρίων Κρέλ και Φανερίστερ Ρόι και λαμβάνοντας υπόψη και τα σχόλια τα οποία έγιναν σε μια προσθήκη που κάνει στο άρθρο 4 παράγραφο 4 ο κύριος Φανίστερ Ρόι ε, στην τροπολογία 19 πιο συγκεκριμένα και όπου εξηγείται γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η προσθήκη νομίζω ότι συνοψίζει πάρα πολύ καλά το ρόλο των ε, τοπικών και περιφερειακών αρχών και τις απόψεις τους. Λέγεται ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η αρχή της συμμετοχής και της εταιρικής σχέσης. Διότι αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι επίσης ε, σημαντικό η όλη αρχή της εταιρικής σχέσης να ε, αναφέρεται και στον κώδικα διοντολογίας. Αυτό που θέλουμε λοιπόν είναι ένα σαφή ορισμό του τι ακριβώς είναι η εταίροι και πώς θα πρέπει να συμμετέχουν οι διάφοροι εταίροι στην πολιτική διαδικασία. Αυτό λοιπόν που επιθυμούμε να επισημάνουμε εμείς από πλευράς τοπικού και περιφερειακού επίπεδου είναι ότι οι δημόσιες αρχές, οι τοπικές και οι περιφερειακές θα πρέπει να θεωρούνται ισότιμοι εταίροι και όχι απλώς ομάδες συμφερόντων ή κάποιες άλλες οργανώσεις. Εμείς είμαστε πεπισμένοι ότι η επιτυχία του προγράμματος εξαρτάται από τη συμμετοχή όλων των εταίρων. Αλλά αναγνωρίζουμε επίσης πόσο σημαντικό είναι να έχουν ιδιαίτερο ρόλο οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, δεδομένως και της νομισμότητας που διαθέτουμε, διότι είμαστε ερετοί, εκλεγόμαστε από, τους, από το λαό και έχουμε λοιπόν ευθύνη και απέναντί τους. επιπλέον είμαστε υπεύθυνοι για πάρα πολλές ε, πτυχές της ε, ζωής και δεν έχουμε μόνο οικονομικές ευθύνες. Σας έχουμε διανύμει τις προτάσεις μας ε, και τις τροποποίησεις που προτείνουμε και θα ήθελα να σταθώ στο άρθρο 5 σημείο 1 εκεί πραγματικά θα θέλαμε να επισημανθεί ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές με τα κράτη-μέλη βεβαίως από κοινού θα πρέπει να είναι αρμόδιες για να οργανώσουν τις εταιρικέ σχέσεις ώστε οι τοπικές και περιφερειακές αρχές να θεωρούνται πραγματικοί εταίροι και όχι απλώς ομάδες συμφερόντων ή οργανώσεις ε, με συγκεκριμένα συμφέροντα. Στον κώδικα θεοντολογίας λέμε ότι αυτό που επιθυμούμε είναι να οριστεί σαφώς ε, τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο εταιρική σχέση. Διότι ελοχεύει ο κίνδυνος, εάν ε, δεν είμαστε ασαφείς, να υπάρχουν προβλήματα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και ιδίως στις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών, εάν δεν είναι σαφές ε, τι ακριβώς εννοούμε όταν περιγράφουμε ε, την ε, εταιρική σχέση. Και σε ευχαριστώ λοιπόν για άλλη μια φορά που μας προσκαλέσατε σε αυτή τη συνεδρίαση και θα σας διανύμουμε και όλα τα σημεία στα οποία αναφέρθηκα. Ευχαριστούμε κυρία Γκούναρσον και τώρα θα ήθελα εξ ονόμως του του κύριου Σίτης να δώσω το λόγο στον κύριο Πολ Τίσλεϊ. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να ευχαριστώ την Επιτροπή σας ε, για την πρόσκληση που μας ε, απέφθηνε να σας μιλήσουμε. Ονομάζομαι Πολ Τίλσλι και είμαι ο δήμαρχος, πρόεδρος μάλλον του Δημοτικού Συμβουλίου του, της πόλης του Birmingham, η οποία έχει δεχθεί σημαντικό ποσό από τον κοινοτικό προϋπολογισμό με σημαντικές ε, ε συνέπειες και αντίκτυπο στην ε, μεταμόρφωση της πόλης μας. Έχουμε ωστόσο σημειώσει σημαντικές ε, ε, εξελίξεις, δυσμενείς δυστυχώς, με σημαντική ε, με σημαντικό αντίκτυπο της κρίσης, ανεργία και κίνδυνο για τους νέους μας. Χωρίς τις κοινωτικές λοιπόν επενδύσεις τα τελευταία 25 χρόνια, το Birmingham θα ήταν μια πόλη όπως το Detroit. Και δεν ομιλώ μόνο για μια πόλη αυτή τη στιγμή, γιατί εκπροσωπώ τη Eurocities. Το δίκτυο δηλαδή των 140 κύριων αστικών κέντρων της Ευρώπης που προσφέρει πολιτική πλατφόρμα και μας επιτρέπει να συζητούμε, να μιλάμε σε επίπεδο ευρωπαϊκό με μία και φωνή. Οι προτάσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αστική διάσταση της πολιτικής συνοχής έχουν στηθεί του τελευταίου έξι μήνε. Σήμερα θα ήθελα συγκεκριμένα να αναφερθώ στι προτινόμενες νέε λύσει, τα νέα μέσα από την οπτική γωνία των πολεών μα των αστικών μας κέντρων. Θα ήθελα ωστόσο ε, πριν το πράξω αυτό να υπογραμμίσω ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, ένα θεμελιώδε ε, ζήτημα, ότι δηλαδή τα μέσα αυτά θα είναι αποτελεσματικά πλήρω μόνο εφόσον η διακυβέρνηση εξασφαλιστεί κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο και θα πρέπει οι κύριε πόλει, τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα, να εμπλακούν απευθεία στι εθνικέ διαδικασίε προσδιορισμού των προτεραιοτήτων για τι επενδύσει. Η ε, ενίσχυση λοιπόν του ρόλου των πόλεων ω εκ τούτου είναι κέρια σημασία για τη διασφάλιση αποτελεσματικών αποτελεσματικής πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, συνεπών στρατηγιών και καλύτερης αξιοποίησης των κονδυλίων και έτσι βελτιστοποίηση της περιφερειακής πολιτικής που διαφορετικά δεν θα εξασφαλιστεί. Δεν θα εξασφαλιστεί. Επιτρέψτε μου τώρα να αναφερθώ στην διελκυστίνδα για την χρηματοδότηση των πόλεων. Θα γνωρίζετε ασφαλώ πολύ καλά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια ελάχιστη διάθεση χορήγηση 5% για ολοκληρωμένη βιώσιμη ανάπτυξη αστικών κέντρων. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει 5% για τις πόλεις, αλλά ελάχιστο ποσό για ολοκληρωμένες ε, εδαφικές επενδύσεις. Και με 75% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ασφαλώς, τα αστικά κέντρα αξίζουν ένα μεγαλύτερο ποσοστό ε, μερίδιο από τις επενδύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο ένα 5% πράγμα το οποίο θα ε, εξασφάλιζε, θα ε, έδινε νέα όθηση σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, εάν εξασφαλιζόταν και θα μας βοηθούσε, θα βοηθούσε τις πόλεις περιφέρειες αυτές ε, να αντιμετωπίσουν προβλήματα που έχουν. Αλλά θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι το 5% αποτελεί μόνο ένα ελάχιστο επίπεδο Εάν όλα τα κράτη-μέρη δηλαδή επιβάλλουν αυτό το ελάχιστο ποσοστό, ή τα αστικά κέντρα θα ε, χάσουν ε, την ευκαιρία να συμμετάσχουν ε, στο τρέχο, στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ρητά να απαιτεί μια ατζέντα για τα αστικά κέντρα για την Ευρώπη. Χρειάζεται σαφής προϋπόθεση τα κράτη-μέλη να μην μειώσουν τη συνολική χρηματοδότηση, χρειάζεται δηλαδή μια σαφέστερη αστική διάσταση σε όλα τα προγράμματα. Και έτσι έρχομαι στο νέο μέσον που είναι γνωστό με τον τίτλο «Ολοκληρωμένοι συνδεφικές επενδύσεις», Integrated Territorial Investments, ITI ε, δηλαδή, που θεωρούμε εμείς στο Eurosys ότι είναι ένα θετικό ε, μέσο ε, για τρεις λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί δίνει έμφαση και ορατότητα σε ολοκληρωμένες και βιώσιμες αστικές ε, δυνατότητες ανάπτυξης. Δεύτερον γιατί προσφέρει την ευελιξία σε γεωγραφικό επίπεδο αλλά και στον προγραμματισμό και την εκτέλεση των κονδυλίων που επιτρέπουν και την ανάπτυξη των οικής σχέσης μέσα στην πόλη, τη, σχέση, τη βελτίωση της σχέσης μεταξύ πόλης περιφέρειας και αστικού κέντρου υπαίθρου σε συνεργατικό επίπεδο και τρίτον γιατί αποτελεί ένα μέσον, μια ευκαιρία οι πόλεις να αναλάβουν τη διαχείριση και την υλοποίηση ευρωπαϊκών επενδύσεων. Η διάθεση λοιπόν, η εκχώρηση της διαχείρισης αυτών των ε, κονδυλίων ε, είναι πάρα πολύ σημαντική. Αποτελεί ως εκ τούτου ένα μέσον και ένα σημαντικό βήμα προόδου και γι' αυτό δεν δεχόμαστε το μάλλον ε, ελαφρά την καρδία προβαλλόμενο επιχείρημα ότι τα αστικά κέντρα δεν έχουν την ικανότητα, το δυναμικό δηλαδή, ότι ε, δεν μπορούν να εκτελέσουν τα έργα αυτά. Σας διαβεβαιώνω ότι υπάρχουν πολλές πόλεις που θα τα καταφέρουν, που είναι έτοιμες, που είναι διατεθειμένες να αναλάβουν ηγετική ε, ηγετικό ρόλο σε εταιρική σχέση με, άλλες, με άλλους φορείς σε τοπικό επίπεδο και ξεκάθαρα μπορώ επίσης να σας πω ότι οι πόλεις και οι τοπικές αρχές έχουν αναπτύξει και έχουν ηγηθεί εδαφικών εταιρικών σχέσεων για δεκαετίες, ως αυτού μια τέτοια προσέγγιση δεν θα ήταν για μας ε, κενός τόπος. Ε, επίσης, θα πρέπει να υπάρχει μια σαφής υποχρέωση ε, για τη διαχείριση, για την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων ITI, των εταιρικών σχέσεων μάλλον ITI στις πόλεις και να έχετε δυνατότητα κάθε πόλη να δεχθεί ή να απορρίψει μια τέτοια πρόταση συνεργασίας. Είναι επίσης πολύ σημαντικό η διαχείριση να επιτρέψει την ανάπτυξη και το δυναμικό που θα φέρει την Ευρώπη του 2020 κατά τρόπο απτό, γιατί δεν είναι σαφές ακόμη το κατά πόσον αυτό θα ε, καταστεί δυνατόν ή πώς θα καταστεί δυνατόν. Ιδιαίτερα υποστηρίζουμε την ιδέα για ένα κατάλογο πόλεων που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την χρηματοδότηση μέσα σε ε, στο πλαίσιο ολοκληρωμένων βιώσιμων ε, αστικών ε, επενδύσεων για την ανάπτυξη. Με ένα τέτοιο λοιπόν κατάλογο οι εταιρικέ συμβάσεις στα λειτουργικά προγράμματα θα μπορούν να βοηθήσουν στην ανάθεση αυτών των ε, επενδύσεων για την ανάπτυξη των περιοχών. Πρέπει όμως και τα κράτη-μέλη σε συνεργασία με τις κυρίες τους πόλεις να αναπτύξουν σαφείς και διαφανείς διαδικασίες και κριτήρια επιλογής για τον κατάλογο αυτό και θα πρέπει να λογοδοτούν βεβαίως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα κράτη-μέλη για τις επιλογές τους. Ο κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει και λειτουργικά και αστικές περιοχές που σε πολλές περιπτώσεις, σε πολλά κράτη-μέλη μπορεί να εκπροσωπούνται από την ε, Μητροπολιτική Πόλη και επίσης σε σχέση με την πλατφόρμα ανάπτυξης των αστικών κέντρων. Πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να προσφέρει προσθέμενη αξία εφόσον διευκολύνει απευθεία διάλογο μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Πόλων σε ολοκληρωμένη ε, βιώσιμη αστική ανάπτυξη, μια πλατφόρμα δηλαδή που μπορεί να βοηθήσει τις πόλεις η μία να διδαχθεί από την εμπειρία της άλλης, να αξιοποιήσουν νέα μέσα, να αναπτύξουν νέο δυναμικό. Αλλά για να προαχθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση πραγματικά χρειαζόμαστε και κάτι περισσότερο από την πλατφόρμα των ανταλλαγών αυτών. Χρειαζόμαστε δηλαδή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη. Πρέπει και οι τρεις να συμφωνήσουν σε ένα νέο τρόπο εργασίας, σε μια νέα μέθοδο εργασίας, μια πραγματικά φιλόδοξη ε, ατζέντα, ένα νέο πρόγραμμα φιλόδοξο για τα αστικά κέντρα που θα σήμαινε και οι πόλεις να, να συμμετάσχουν πιο ενεργά και απευθεία στη διατύπωση και τη διαχείριση των λειτουργικών προγραμμάτων και ε, όλοι οι αρμόδιοι επίτροποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αναζητήσουν ευκαιρίες διαλόγου με δημάρχους όταν επισκέφτονται κράτη-μέλη και τρίτον να ξεκινήσει μια σειρά δραστηριοτήτων για τα αστικά κέντρα, αντίστοιχη με αυτή των ανοιχτών θυρών σε συνεργασία με την Επιτροπή των Περιφερειών. Έτσι λοιπόν πιστεύουμε ότι θα πρέπει για τέσσερα βασικά σημεία να ε, συμμετέχουν απευθεία οι πόλει στι εταιρικέ σχέσει που προσδιορίζουν προτεραιότητε, ε, με τρόπο σαφή όμω να οριστεί αυτό στο άρθρο 5 του Γενικού Κανονισμού. Δεύτερον, θα πρέπει να εφαρμοστεί μια σαφή αστική προτεραιότητα για όλε τι ε, προτεραιότητε επενδύσεων του άρθρου 5 του ε, Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εκχωρίουν ε, την χρηματοδότηση σε επίπεδο πόλεων και λειτουργικών αστικών κέντρων έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται πιο συγκεκριμένα οι τοπικές προκλήσεις. Σε τελευταία ανάλυση οι πόλεις είναι εκείνες που ε, αποτελούν και θα αποτελούν και στο μέλλον το κλειδί για την υλοποίηση της εδαφικής συνοχής και των στόχων της Ευρώπης του 2024. θα πρέπει να υπάρχει ρητή και διαφανής επιλογή των πόλεων για την ε, ε, ξεκάθαρη μάλλον και διαφανής επιλογή των πόλεων για την εκχώρηση των κονδυλίων ε, που στήριζονται σε εθνικές διαδικασίες και κριτήρια αναπτυσσόμενα σε συνεργασία με τις πόλεις, όπως, θα πρέπει μάλλον προκύπτει ξεκάθαρα από το άρθρο 7 του κανονισμού για την περιφερειακή ανάπτυξη. Με αυτή τη... Και θα ήθελα κλείνοντα να σας πω ότι η ταχύτητα των αλλαγών στην Ευρώπη, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές αλλαγές είναι τεράστια. Η ταχύτητα των αλλαγών είναι τεράστια. Έχουμε μπει στην αφετηρία μιας νέας επταετούς περίοδου όπου οι πόλεις και οι πολίτες θα αποτελέσουν το επίκεντρο των αλλαγών αυτών, το να προσφερθούν λοιπόν, το να διατεθούν τα μέσα και τα εργαλεία ε, σε εμάς θα σήμαινε ότι είμαστε σε θέση να, ότι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τις αλλαγές αυτές σε τρόπο και βιώσιμο και διαρκή. Η ευκαιρία δεν είναι ε, δεν είναι μια ευκαιρία που μπορεί να χαθεί. Δεν πρέπει να χαθεί η ευκαιρία αυτή. Διαφορετικά κινδυνεύουμε να χάσουμε και την ευκαιρία του 2020. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ε, ήταν πολύ σημαντική αυτή η έκκληση και προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και έχουμε και υποχρέωση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Θα ακούσουμε τους ειδικούς μας ηγητές, όχι μόνο βέβαια, την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε και ένα προσκεκλημένο από τη Βουλή της Τοσκάνης. Θα του δώσουμε το λόγο να λάβει μέρο στη συζήτηση. Πάντως όσοι θέλετε το λόγο, παρακαλώ να το δηλώσετε για να μπορέσουμε να δούμε πόσο χρόνο δικαιούται ο καθένας. Θα ξεκινήσω από τους συζητητές για το γενικό κανονισμό. Φαντάζομαι ο Λαμπέρ θα είναι ο πρώτος που θα λάβει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ ευχαριστώ να λάβω το λόγο και να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους μας για το πνεύμα κυρίως των ομιλιών τους που ήταν πολύ φιλόδοξο και για την ετοιμότητα και προθυμία τους να βελτιώσουν τις τρέχουσες πρακτικές γιατί δεν δημιουργούμε κάτι καινούριο, απλώς αξιοποιούμε κάτι που έχει προταθεί εδώ και χρόνια για αποκεντρωμένη διακυβέρνηση και εταιρική σχέση. Θέλουμε καλύτερη συνεργασία και καλύτερο συντονισμό και καλύτερη στοχοθέτηση για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις ε, που θα αντιμετωπίσουμε μέχρι το 2020. Από τη σημερινή συζήτηση πάντως, το πιο σημαντικό σημείο που ανέκυψε είναι ότι Αυτά τα ζητήματα απασχολούν ε, όλα τα κράτη-μέλη, γιατί πραγματικά οι περιφέρειες είναι οι εταίροι των ε, κεντρικών κυβερνήσεων και σημαντικό είναι να συνεχιστούν οι συζητήσεις και εκεί, γιατί με την κρίση κάθε δύο-τρεις μήνες προκύπτει και μια νέα πρόταση, ένα νέο σχέδιο δράσης. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα υπάρχοντα μέσα και τους βασικούς χρηματοπιστωτικούς και δημοσιονομικούς κανονισμούς για να χρηματοδοτήσουμε τις πολιτικές μας. Πάντως, χαίρομαι για το πνεύμα που επικράτησε, το πνεύμα του ενθουσιασμού και στην Επιτροπή των Περιφερειών, που ασχολείται και αυτή με το θέμα και συμπνέει με τα δικά μας σχόλια. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αρχή της εταιρικότητας, είναι σημαντικό και έχουμε ήδη ένα κείμενο, θα προσπαθήσουμε να εκλεπτύνουμε κάπως αυτή την έννοια και να τροποποιήσουμε τη διατύπωση του άρθρου 1 για να διευκολύνουμε την εταιρική σχέση με, τους, με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Επίσης, θέλουμε και ένα είδος συνεννόησης, συν, ομοφωνίας για την, συνένεση για την εταιρική σχέση μεταξύ των διαφόρων εταίρων στην προκαταρκτική φάση του σχεδιασμού για να αποφύγουμε μια επανεθνικοποίηση της πολιτικής συνοχής και εκεί θα διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο και το Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη σας και θα επεξεργαστούμε ιδιαίτερα αυτό το σημείο. Ένα άλλο θέμα που είναι πολύ ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου και για το οποίο θα θέσω και μία ερώτηση είναι το εξής. Τι γίνεται με αυτή την ε, ευφύ εξειδίκευση των διαφόρων περιφερειών. Ποια θα είναι η συμβολή τους, πώς ε, θα επιταχύνουμε το δρόμο προς την αριστεία. Με την έρευνα, με την καινοτομία, σίγουρα με τις υποδομές, είναι τομείς προτεραιότητας. Έχουμε επίσης την οικονομία που θα πρέπει να στηρίζεται στη γνώση. Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αυτά τα σημεία. Και το θέμα της ε, εδαφικής συνοχής επίσης είναι πολύ σημαντικό και τονίστηκε. Αυτά τα θέματα θα ήθελα να τα εξετάσουμε και σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο και όχι μόνο σε ευρωπαϊκό. Βέβαια, όταν επικεντρωνόμαστε σε ένα τομέα μόνο, μπορούμε να έχουμε καλύτερο συντονισμό μεταξύ των περιφερειών και της γνώσης των περιφερειών. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Και αυτό το, το σχέδιο να το μεταλα, μεταλαμπαδεύσουμε και στις, στην περιφερειακή συνεργασία, διαπεριφερειακή συνεργασία. τι γίνεται με τις μειονεκτικές περιοχές, λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές. Προσπαθούμε να τους ε, να τις υποχρεώσουμε να επενδύσουν κάποια κονδύλια από τον προϋπολογισμό τους σε συνεργασία με τις ε, πιο ανεπτυγμένες, πιο ισχυρές περιφέρειες. Έτσι θα έχουμε μια αλληλοβοήθεια μεταξύ των περιφερειών, ώστε όλες ε, οι περιφέρειες να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις βέλτιστες πρακτικές, ε, τη γνώση και χρησιμοποιώντας την καινοτομία να προωθήσουν την κατάρτιση, την επιχειρηματικότητα και να δημιουργήσουν και θέσεις απασχόλησης. Αυτό είναι το δικό μου όραμα για την Ευρώπη του 2020. Και τέτοιου είδους ανάπτυξη επιδιώκουμε. Εσείς τι γνώμη έχετε γι' αυτό. Γιατί έτσι νομίζω θα μπορέσουμε να έχουμε και συνέργεια στα πλαίσια ε, του ερευνητικού προγράμματος ε, για το 2020 και συνέργεια μεταξύ του ερευνητικού προγράμματος και του περιφερειακού προγράμματος. Αυτά και περιμένω τις απόψεις. Η Κωνσταντζα Κρέλ, που είναι επίση εισηγήτρια, συνεισηγήτρια για το Γενικό Κανονισμό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Οι συγγετικέ παραβάσει ε, μας δίνουν την εντύπωση ότι όντω έχουμε πολύ καλή συνεργασία ήδη εδώ και καιρό. Τα πιο σημαντικά σημεία τα οποία εξετέθησαν τα έχουμε ήδη σε μεγάλο βαθμό ενσωματώσει στην έκθεσή μας και μπορούμε να περιμένουμε νομίζω και ευρύτερη η πλειοψηφία που θα υποστηρίξει και σε επίπεδο επιτροπή και σε επίπεδο λομέλεια στην έκθεση αυτή. Θα ήθελα σε κάποια σημεία μόνο να επισέλθω. Το ένα αφορά την, ε, τους ε, μακροοικονομικούς όρους θα πρέπει πιστεύω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταστήσουμε σαφές ότι οι μακροοικονομικές προϋποθέσεις και η κατάσταση δημοσιονομική στο ιστορικό των κρατών μελών δεν έχει καμία σχέση με την περιφερειακή πολιτική. Είναι άσχετα μεταξύ του. Βεβαίω είναι απαραίτητα και τα δύο, αλλά δεν μπορούμε την πολιτική συνοχή τη περιφέρεια να την υπαγάγουμε στην ε, εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα δημοσιονομικά του οι εθνικέ κυβέρνησει. Πρέπει να βρούμε ένα διαφορετικό τρόπο, πιστεύω, και γι' αυτό νομίζω προτείνουμε ε, και πολύ σωστά τη διαγραφή του άρθρου 21. Ξέρω ότι δεν θα συμφωνήσουν οι πάντε, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα εξασφαλιστεί ευρύτερη πλειοψηφία σε Κοινοβουλίου, πάντω στην Επιτροπή μα, για τη του άρθρου αυτού. Αυτό που δεν θα θέλαμε είναι το μέσον το οποίο υφίσταται ήδη μέσα από το Ταμείο Συνοχής και επιτρέπει την ανάληψη μέτρων να διαγραφεί. Αυτό θέλουμε να διατηρηθεί γιατί έχει σημασία και το Ταμείο Συνοχής έχει ε, εφευρεθεί για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν προς την νομισματική ένωση, προς το ευρώ. Εξ εκ τούτου λοιπόν η συνοχή εξαρτάται πράγματι από την ε, πραγματική προσπάθεια που θα αναπτύξουν τα κράτη-μέλη με, με στόχο την εξυπηρέτηση, την τήρηση των κριτηρίων ε, του ευρώ και της νομισματικής Ένωση. Αυτό είναι ο στόχο του, αλλά δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αποτελέσει ένα μέσον εκφοβισμού των κρατών μελών και να τα υποχρεώνει να ακολουθούν μια συγκεκριμένη δημοσιονομική πολιτική με, με φόβητρο την ε, διακοπή τη χρηματοδότηση από την πολιτική συνοχή. Γι' αυτό λοιπόν και εμεί είμαστε δραστικά κατά ε, του άρθρου 21 και θέλουμε τη διαγραφή του. Επίσης, Πιστεύουμε και συμφωνούμε στην Επιτροπή μας ότι θα πρέπει η ανάπτυξη των αστικών κέντρων να αποτελέσει επίκεντρο της ε, πολιτικής της συνοχής, όχι μόνο γιατί εκπροσωπούν τα αστικά κέντρα το 75% των πολιτών, ζουν σε αυτά δηλαδή 75% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και γιατί η πολιτική της συνοχής μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από τα αστικά κέντρα, με την βελτίωση φερρυπίν της αποτελεσματικότητας της ε, χρήση ενέργειας, με τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Όλα αυτά είναι στόχοι που υλοποιούνται μέσα από τα αστικά αστικά κέντρα και γι' αυτό θέλουμε να είναι το ελάχιστο αυτό όριο ένα όντως ελάχιστο όριο και να επιδιώκουμε γενικότερα υψηλότερου στόχου για συμμετοχή των αστικών κέντρων στην πολιτική αυτή. Και ω εκ τούτου θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να καθίσατε σαφέ μέσα από το κείμενο ότι τα αστικά κέντρα και η ανάπτυξή του έχει ιδιαίτερη σημασία για μα και για την υλοποίηση της πολιτικής συνοχής. Ε, ωστόσο υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες και γι' αυτό θα ήθελα να διατυπώσω και την σχετική συμπληρωματική ερώτηση. Εάν έχει νόημα ένα επιπλέον ε, φόρουμ για τις ανταλλαγές ε, απόψεων μεταξύ των πόλεων. Η δική σας η ένωση, η σας οι δικές σας πλατφόρμες δεν αποτελούν αυτή την ε, βάση ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών. Χρειάζεται πραγματικά να δώσουμε νέες δομές, ε, χρειάζεται πράγματι να περάσει αυτό μέσα, ε, να, περνούν μέσα από μια νέα τέτοια ε, οργάνωση ή προτάσεις για τα καλύτερα σχέδια για τις πόλεις, τα αστικά κέντρα κτλ. Και επίσης πιστεύω ότι ένας ενδεικτικός πίνακας για τα αστικά κέντρα στην αρχή της ε, διαδικασίας θα μπορούσε να αποτελέσει παράγοντα περιορισμού της ευελιξίας που θα είχαμε διαφορετικά. Δηλαδή θα έλεγα καλύτερα να προσδιορίσουν τα κράτη-μέλη τι εννοούν ως αστικό κέντρο ή να αφήσουν να δούμε τι σημαίνει λειτουργικό αστικό κέντρο ή λειτουργική περιφέρεια με κάποια κριτήρια προκαταβολικά και όχι να πούνε ε, ε, εξ αρχής ποια είναι τα αστικά κέντρα στα οποία στοχεύουν. Πάντως δική μας δουλειά δεν θα πρέπει να είναι. Δεν ξέρω εσείς τι, πιστεύετε σε αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι δουλειά μας να προσδιορίζουμε κριτήρια δηλαδή. Πέραν αυτών των βασικών. Να μην, δηλαδή δεν θα πρέπει να ορίσουμε καταλόγους που ενδεχομένως να οδηγήσουν και σε αντιπαραθέσεις και εντάσεις στο εσωτερικό κρατών μελών άμα ε, στέλνει στους κατάλογους, θα έχουμε πολύ περιορισμένες δυνατότητες να τον τροποποιήσουμε στην πορεία του προγράμματος. Γι' αυτό η δική μας επιλογή είναι πιο ε, αποτελεσματική, πιστεύω, και για τις περιφέρειες και για τα αστικά κέντρα. Θα ήθελα να ακούσω όμως τις δικές σας απόψεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους προσκεκλημένους, τους εκπροσώπους των τοπικών και περιφερειακών αρχών, όχι μόνο για την παρουσία τους, αλλά και για τα έγγραφα που μας έδωσαν. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα σημεία που ήταν κοινά στοιχεία και των τεσσάρων ομιλιών. Παρόλο που υπάρχουν ε, φυσικά και μερικά στοιχεία που λογικό είναι να είναι διαφορετικά μεταξύ των ε, διαφορών οργανώσεων γιατί κάθε οργάνωση ε, εκπροσωπεί διαφορετικούς φορείς. Είναι σημαντικό να υπάρχουν και κάποιες διαφορές. Ο πρόεδρος της διάσκεψης απομακρυσμένων περιφερειών μίλησε για ορισμένα σημεία που είναι κοινά σημεία σε όλους, αλλά υπάρχουν και μερικά διαφορετικά σημεία. Είναι λογικό φυσικά, είναι φυσιολογικό, γιατί αν ήταν απόλυτη η των απόψεων και των τεσσάρων οργανώσεων, θα χρειαζόμασταν τέσσερι διαφορετικέ οργανώσει, θα αρκούσε και μία, αν υπήρχε πλήρη σύμπνοια και ομοφωνία. Θα ήθελα να αναφερθώ στα πιο θεμελιώδη ζητήματα. Το πρώτο θέμα που αναφέρεται σε όλα τα έγγραφα και στις ομιλίες ε, των ε, προσκεκλημένων είναι το θέμα της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και κυρίως το θέμα της εταιρικότητας, της εταιρικής σχέσης και το θέμα του κώδικα συμπεριφοράς, του διοντολογικού κώδικα. Και σε αυτό αναφέρεται και η ερώτησή μου. Ε, συνεχίζονται οι συζητήσεις μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτό το λεγόμενο κώδικα συμπεριφοράς. Κατά τη γνώμη σας, ένας τέτοιος κώδικας θα πρέπει να έχει πανευρωπαϊκό χαρακτήρα, θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκός κώδικας ή να αποτελέσει το αντικείμενο των διαπραγματεύσεων μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών αρχών και των εταίρων τους. Είναι πολύ σημαντικό. Θα έχουμε ένα μοντέλο που θα ισχύει για όλες τις, δια... τις διαφορετικές μορφές εταιρικότητας. Γιατί έχουμε τα θέματα των εταιρικών συμβάσεων, των συμβάσεων εταιρική σχέσης και ποιος θα είναι ο εταίρος αυτός, πώς θα ορίσουμε τον εταίρο, ποιος θα προσκαλείται στις εργασίες για την εταιρική αυτή σύμβαση. Πώς θα αντιμετωπίζεται αυτός ο εταίρος, ποιες θα είναι οι αναλογίες μεταξύ των τοπικών περιφερειακών εταίρων και των λοιπών εταίρων ή των, των μη κυβερνητικών οργανώσεων ή των ε, κυβερνήσεων. Είναι πολύ ευαίσθητο αυτό το σημείο, πολύ λεπτό, γιατί θα καθορίσει και τον προγραμματισμό των, των κονδυλίων, της κατανομής των κονδυλίων σε ε, κρατικό επίπεδο. Λοιπόν, αυτός ο ορισμός θα πρέπει να γίνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ή να το αφήσουμε στα κράτη-μέλη να λαμβάνουν αυτά την απόφαση για τις εταιρικές σχέσεις. Ό,τι αφορά τώρα τις συμβάσεις εταιρικής σχέσης, ε, και εδώ έχουμε πολλά και διάφορα σημεία. Ένα από αυτά είναι αυτός ο περίφημος κατάλογος ε, των ε, συνεδρίων. Μία πρόταση που θα στηρίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι υπέρ ε, του καταλόγου των πόλεων, αλλά το καταλόγου των κριτηρίων που θα πρέπει να καταρτιστούν σε εθνικό επίπεδο. Γιατί δεν υπάρχει ένα ενιαίο κριτήριο που μπορεί να ισχύσει πανευρωπαϊκά τα κριτήρια για το περίφημο αυτό 5% του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι πολύ σημαντικό θέμα. Οπότε ο κατάλογος, κατά τη γνώμη μας, θα πρέπει, ο κατάλογος των πόλων θα πρέπει κατά τη γνώμη μας να καταργηθεί. στον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, για, το οποίο, για τον οποίο είμαι εισηγητής, προτείνω την κατάργηση και των πλατφορμών των πόλεων και πιστεύω ότι θα πρέπει να προβλέψουμε άλλους μηχανισμούς επιτήρησης και αξιολόγησης. Υπάρχει και ένα θέμα Όλο αυτό το πακέτο μάλλον αφορά τις, ε, τις σχέσεις εταιρικότητας και τις συμβάσεις εταιρικής σχέσης. Ένα άλλο ζήτημα που αφορά το ενιαίο στρατηγικό πλαίσιο. Ποιο θα πρέπει να είναι το νομικό καθεστώς αυτού του στρατηγικού πλαισίου για το ζήτημα αυτό έχουμε και την πιο πρόσφατη πρόταση των εισηγητών μας, των συνεισηγητών, που μιλούν για κοινό στρατηγικό πλαίσιο. Θα πρέπει να είναι νομοθετικό αυτό, νομοθετική αυτή η πράξη, κατεξουσιοδότηση πράξη. Τι μορφή θα πρέπει να λάβει, ποιος θα πρέπει να είναι ο νομικός χαρακτήρας αυτού του κοινού στρατηγικού πλαισίου γιατί αφορά τις ε, δράσεις κλειδιά και τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων ταμείων γιατί δημιουργείται μια αμφιβολία για το νομικό καθεστώς και θα πρέπει οπωσδήποτε να διασκεδαστεί. Ένα άλλο σημαντικό θέμα που προέκυψε από τις ομιλίες σας είναι ε, ένα ζήτημα που προέκυψε στο ΦΕΝΤΕΡ, το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, για τις ε, επενδύσεις των πλέον ανεπτυγμένων περιφερειών και ένα θέμα που σχετίζεται και με τη θεματική συγκέντρωση. Και δώσω ε, συζητήσεις για το ζήτημα αυτό εγώ θα πρότεινα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την κατάργηση του σχετικού περιορισμού. Θα δούμε αν θα ευοδοθεί αυτή η πρόταση. Εγώ θα προτείνω την κατάργηση του περιορισμού σε ό,τι αφορά τις υποδομές των πλέον ανεπτυγμένων ε, περιφερειών. Άλλωστε η σημερινή κρίση νομίζω συνηγορεί υπέρ της κατάργησης του σχετικού περιορισμού του σχετικού σημείου. Θα ήθελα ανακεφαλαιώνοντας ε, να σας ε, θέσω την ερώτηση ε, κυρίως ε, για τον κώδικα συμπεριφοράς. Σε ποιο επίπεδο θα πρέπει να προσδιοριστεί αυτός ο κώδικας συμπεριφοράς ε, και ποια θα πρέπει να είναι η λύση που θα πρέπει να δώσουμε για αυτόν τον κώδικα συμπεριφοράς. Ευχαριστώ. Τώρα να κάνω μια γενική παρατήρηση. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι πάρα πολύ μεγάλος ο κατάλογος. Σας παρακαλώ, προσπαθήστε λοιπόν να κάνετε τις παρατηρήσεις σας εντός τριών λεπτών και επικεντρωθείτε μόνον στα όσα μας παρουσίασαν οι φίλοι από τις ε, ε ενώσεις. Ε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ε, καλωσορίσω και τους εκπροσώπους των πόλων και των περιφερειών που έχουμε εδώ προσκεκλημένους και να ε, τους ευχαριστήσω για τη συμμετοχή τους εδώ στη συζήτηση. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει και στην εθνική, στον εθνικό θυμόσο διάλογο που έχει ήδη ξεκινήσει να συμμετάσχουν προδραστήρια. Διαπιστώνουμε ότι οι στόχοι για την πολιτική της συμμετοχής με ε, με τα κριτήρια της Ευρώπης του 2020 θα έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία. Ακούμε από διάφορες περιφέρειες ότι απαιτείται απασχόληση ανάπτυξη με μέσα της πολιτικής της συνοχής να υποστηριχθούν δεδομένης της οικονομικής κρίσης και βλέπουμε με ανησυχία ότι τα κράτη εκείνα τα οποία θα έπρεπε να επωφελούνται περισσότερο προ τα ποσά τουλάχιστον από την πολιτική συνοχή είναι ακριβώ εκείνα τα οποία δεν είναι σε θέση να αξιοποιήσουν στο βαθμό τουλάχιστον που απαιτείται τα κονδύλια και να τα απορροφήσουν και σε αυτό χρειάζονται νέα μέσα χρηματοδότησης. Έτσι λοιπόν και όπως είπαν και οι συνάδελφοι ήδη, διατυπώνω ένα ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι διαπραγματεύσεις για τις ε, συμφωνίες εταιρικής σχέσης σε ποιο βαθμό έχουν προχωρήσει. Έπρεπε να είχαν ξεκινήσει το Μάρτιο ε, φέτος επαφές μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κρατών μελών, εταιρικέ ε, συμφωνίες εταιρικής σχέσης οι οποίες θα έπρεπε να έχουν συναυθεί με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Αλλά σε αυτές οι περιφέρειες έχουν συμμετάσχει, γιατί αυτές εκπροσωπούν την περιφέρεια, έχουν εκπροσώπηση επιδοκρατών μελών ε, ή φροντίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Περιφερειακή Διάσταση να λαμβάνεται υπόψη για τα αστικά κέντρα και το ελάχιστο ε, ποσοστό του 5% για τη συνολική διάθεση κονδυλίων σε ένα κράτο ε, μέλο. Ε, ακούω πληροφορίε από διαπραγματεύσει μεταξύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διαφορών συνεργατών και εταίρων που είναι αρμόδιοι για την διαμόρφωση των λειτουργικών προγραμμάτων. Το σχόλιο, το 5% των κονδυλίων ε, δεν είναι και τόσο πολλά χρήματα πρώτον. Δεύτερον, ότι είναι διαφορετικέ οι προτεραιότητε, δηλαδή Ευρώπη του 2020 και κυρίω ανάπτυξη και απασχόληση. Και τα αστικά κέντρα μπορούν να αποτελέσουν ένα χώρο ιδιαίτερης ή ιδιάζουσας ανάπτυξης, ενίσχυση καλύτερα, και η συζήτηση την οποία ακούω από την άλλη πλευρά, από πλευρά του Συμβουλίου δηλαδή, δεν δείχνει να διαμορφώνονται συμφωνίες. Βλέπουμε παραδείγματι ότι έχουν συνασπιστεί ορισμένα κράτη σε μια ομάδα που ονομάζεται Friends of Better Spending ε, οι υποστηρικτέ, δηλαδή τη καλύτερη διάθεση των κονδύνων ενώ από την άλλη ω αντίπαλο δέο, ε, έχουμε την ομάδα των Friends of Cohesion, φίλοι τη συνοχή ε, που θέλουν να συνεχιστεί η πολιτική της και να ενισχυθεί η πολιτική τη συνοχή, πράγμα το οποίο βεβαίω εμεί ω αντικείμενο ως κομμάτι τη πολιτική τη περιφερειακή, το βλέπουμε και θέλουμε να παραμείνει η πολιτική συνοχής κομμάτι τη περιφερειακή πολιτική. γι' αυτό λοιπόν μια ερώτηση για του εκπροσώπου των περιοχών εκείνων οι οποίε είναι περιοχές στόχου 2 ανάπτυξη και απασχόληση δηλαδή ε, και ερωτώ πώς τάσσονται σε σχέση με τους, τη στόχευση και τα ποσοστά που προσδιορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 20% δηλαδή ε, μόνο για την ε, μετάβαση 80% ε, για την καινοτομία, την απασχόληση κτλ. Πώς βλέπετε λοιπόν αυτή τη ταξινόμηση στην οποία προβαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Μαρία Ρικογιάν Πέρες. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη για τη μικρή καθυστέρηση. Έπρεπε να κάνω μια παρέμβαση σε μια άλλη επιτροπή. Επομένω δεν ήμουν παρούσα στις ε, παρουσιάσει των εκπροσώπων των πόλων. Ήμουν όμως παρούσα και άκουσα πόσο απαραίτητο είναι τα ταμεία να μπορέσουν να συμπληρωθούν και να προσπαθήσουμε να βρούμε την απαραίτητη αποτελεσματικότητα και το γεγονός ότι οι πόλεις έχουν το μεγαλύτερο ε, ε, δίκτυο, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος του Μπέρμιγχαμ. Προσπαθούμε λοιπόν να εξεύρουμε αποτελεσματικότητα και συνέργεια μεταξύ των ταμείων και να βρούμε και την ε, δυνατότητα να είναι αυτό που πρέπει να είναι. Και είναι πολύ σημαντικό να γίνεται αυτός ο άμεσος διάλογος μεταξύ των τοπικών εκπροσώπων που γνωρίζουν ποιες είναι οι ανάγκες των πολιτών τους ε, και να μπορέσουμε να κάνουμε ενεργές πολιτικές απασχόλησες και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα ταμεία για να δοθούν οι πόροι αλλά ταυτόχρονα και να δοθούν οι δυνατότητες να εξευρεθούν θέσεις εργασίας ιδίως σε καιρό κρίσης όπως είμαστε τώρα. Και φυσικά είμαστε υπέρ της συνέργειας και της συμπληρωματικότητας των ταμείων και ε, να εξεύρουμε πώς μπορούμε να τα βελτιώσουμε. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι ένα σημαντικό παρακλάδι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση, αλλά θα πρέπει να ενισχυθεί. Δεν μπορούμε ε, να ε, το ε, ε στερήσουμε από όλη την ουσία. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να εργαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να βρούμε την κατάλληλη συμπληρωματικότητα και με τις διευκρινήσεις που έκανε η συνάδελφος Κωνσταντς Κρέλ για το ποιο θα πρέπει να είναι το κοινό δημοσιονομικό πλαίσιο, να προσπαθήσουμε να βρούμε αποτελεσματικότητα μέσω διαλόγου. Δεν χρειαζόμαστε νέες πλατφόρμες, αλλά να ενεργοποιήσουμε καλύτερα και να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα αυτές που διαθέσουμε και να προσπαθήσουμε να βρούμε ένα αποτελεσματικό τρόπο προς όφελος των πολιτών που περιμένουν μια απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Ο Αλέν Καντέκ. Merci, Madame la Présidente. Ευχαριστώ. Και εγώ έχω λίγα λόγια επί των παρεμβάσεων των προσκεκλημένων, τους οποίους ευχαριστώ θερμά, τους εκπροσώπους των περιφερειών, για τις παρεμβάσεις τους και για τις προτάσεις τους για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Και χαίρομαι που υπενθυμίστηκε ο σημαντικός ρόλος του Κοινοβουλίου και των βουλευτών σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση αυτής της πολιτικής και ευχαριστώ και την Κωνσταντ και τον Λαμπέρ, τους δύο συνεισηγητές για το έργο τους. Νομίζω ότι είναι, ήταν εύστοχη αυτή η πρόταση για τον ορισμό δύο συνεισηγητών για ένα τόσο σημαντικό έγγραφο του Γενικού Κανονισμού. Και νομίζω ότι ίσω είναι και παράδειγμα προ και για άλλε επιτροπέ αυτό ο διπλό διορισμό εισηγητών. Σε ό,τι αφορά την παρέμβαση του Ζανίβ Λεντριάν, του Προέδρου τη Διάσκεψη Απομακρυσμένων και Θαλάσσιων Περιφερειών, παρόλο που η μακροοικονομική ερεσιμότητα είναι ένα θέμα προσφυλέ για πολλού από εσά, δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να δημιουργήσει αδιέξοδο ή να κολλήσουμε σε αυτό. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω τέτοιο σκοπό. Κάτι που ισχύει και για τη δική, μας, σας περιφέρεια, αλλά και για τις υπόλοιπες, θα πρέπει να συμβάλλουν στην εξυγίανση των δημοσιονομικών τους και να προβλέψουν τις απαραίτητες προσαρμογές. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να το τονίσουμε. Τώρα, περισσότερε ευθύνε ό,τι αφορά την χρησιμοποίηση των κονδυλίων για τις περιφέρειες, αλλά θα πρέπει οι περιφέρειες να αναλάβουν και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από μια τέτοια αύξηση των αρμοδιοτήτων. Και τέλος, ό,τι αφορά την πρόταση του πρόεδρου του ΕΡΠΕΜ, συμφωνώ σε ό,τι αφορά τις τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφορίας που θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα της πολιτικής συνοχής. Σε ό,τι αφορά την παρέμβαση της Μισελ Σαμπάν, Πρόεδρου της Συνέλευσης των Περιφερειών της Ευρώπης, είναι σημαντικό να έχουμε μια θεματική συγκέντρωση σε 11 προτεραιότητες, κάτι που απορρέει από τη Στρατηγική Ευρώπη 2020 και προβληματίζομαι κατά πόσο είναι ε, πρόσφορο το αίτημα των Eurocities σε ό,τι αφορά την ελεύθερη επιλογή αυτή αυτής της συγκέντρωσης. Γιατί ίσως κάτι τέτοιο δημιουργήσει κατακαιρματισμό των κονδυλίων και περιορίσει την προστιθέμενη αξία τους. Προσοχή λοιπόν σε αυτό το αίτημα. Αυτές λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, ήταν οι παρατηρήσεις εκ μέρους μου. Πάντως, το έργο των συνεισηγητών είναι πάρα πολύ αξιόλογο, καταπληκτικό και θα συμβάλλουμε κι εμείς με την υποβολή τροπολογιών. Η ε, κυρία Μαριταρέ Σάντσες Σμιτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω όλους ε, όσοι έλαβαν το λόγο που μας ε, προσέφεραν την πολύ σημαντική του συμβουλή για την επεξεργασία της προσεχούς πολιτικής συνοχής. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι μαζί με το ότι στο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχετε ένα σύμμαχο για φιλόδοξες προτάσεις, για προτάσεις εταιρικέ, συνεργατικές που βλέπω ότι αποτελεί το αίτημα όλων των όσοι έλαβαν τον λόγο. Ιδιαίτερα θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι έχετε δίκιο να απαιτείτε εταιρική σχέση ε, με την δυνατότητα συμμετοχή για κάθε τοπική περιφερειακή αρχή που θα πρέπει να συμμετέχει στο ευρωπαϊκό εγχείρημα που εξυπηρετεί άλλωστε και την ευρωπαϊκή στρατηγική. Και θέλω να υπογραμμίσω ιδιαίτερω ότι μπορεί η πολιτική της συνοχής να είναι πολιτική επενδύσεων στις ε, περιφέρειες στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με προαγωγή του καλύτερου, του, των πιο θετικών στοιχείων τους, θα πρέπει ταυτόχρονα ωστόσο να έχουμε και μια ευρωπαϊκή στρατηγική, μια μακροπρόθεσμη στρατηγική. Οι ευρωπαϊκές επενδύσεις δεν αντιποκαθιστούν τις εθνικές ή περιφερειακές επενδύσεις, υλοποιούν απλώς μια περιφερειακή στρατηγική συνοχής και θα πρέπει να την βελτιώνουν. Θα ήθελα ιδιαίτερα να υπογραμμίσω για τη συνέργεια ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αντιταχθεί στην αρχή της επικουρικότητας όσον αφορά τον προσδορισμό μιας εταιρική σχέσης. Μόνο μπορεί να την υποστηρίξει αυτή την αρχή με ιδιαίτερη έμφαση. Και θα ήθελα σε σχέση με την διατύπωση που προτείνουν οι συντάκτες της εκθέσεως για την εταιρική σχέση να υπογραμμίσω ότι μπορεί να ε, ικανοποιήσει τις προσδοκίες σας πιστεύω γιατί αναφέρει ρητά την εταιρική σχέση, ορίζει ότι θα γίνεται μέσα στο θεσμικό πλαίσιο αλλά στο κατάλληλο εδαφικό επίπεδο ε, και σε συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και των προσδοριστέντων από τα ίδια τα κράτη-μέλη φορέων και στην υλοποίηση και στην, ε, στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση και στην εκτέλεση και θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στις ε, προτάσεις ε, του Ισραήλ των Περιφερειών της Ευρώπης για συμβιβασμούς, για διάθεση για συμβασμό καλύτερα που θα αποέβαινε προς όφελος των πάντων ε, στο στόχο του, της εξασφάλισης επενδύσεων. Αλλά η πραγματική εταιρική σχέση πιστεύω και υπογραμμίζω πρέπει να αποτελεί τον εκτρόνου κάνευ όρο ε, για τους ε, στόχους μας, για το σχεδιασμό μας, για την Ευρώπη του 2020. Και ο κ. Καντέκ, η Ευρώπη απαιτεί και συμμετοχή στη σταθεροποίηση που είναι απαραίτητη για την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Μάνκα. Μάσκα. E, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τους φίλους μας, εκπροσώπους των πόλεων και των περιφερειών. Υπήρξα δήμαρχος ε, μιας ε, πόλης ε, και είμαι και επικεφαλής της περιφέρειας αυτή τη στιγμή και καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι εννοούν. Ζητούν οι περιφέρειες να έχουν αρκετό περιθώριο να λαμβάνουν αποφάσεις για αυτά τα οποία θα δοθούν ως κονδύλια στην αντίστοιχη περιφέρεια. Θα ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα επί τη βάση του οποίου μπορούμε να κάνουμε περαιτέρω συζητήσεις. κάποιες περιφέρειες ε, τοποθετούν πλέον μόνο στα κτίρια και ρωτήθηκε ποια είναι η προστιθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας πω το εξής. Όταν εγώ έγινε επικεφαλής της περιφέρειας ε, πριν από 2,5 χρόνια, ζήτησα να μου δοθεί ένας κατάλογος για όλα τα κτίρια και όλα τα αγαθά που διαθέτει η περιφέρεια. Και διαπίστωσα ότι, για παράδειγμα, στα σχολεία, αν υπάρχουν μεγάλες ενεργειακές απώλειες, ε, και κάνω μια επένδυση σε καλύτερη θερμομόνωση για τα σχολεία, αυτό εξοικονομεί χρήματα τα οποία μπορώ να χρησιμοποιήσω για άλλο σκοπό. Και φυσικά έχει θετικές επιπτώσεις και για το περιβάλλον αποταμιεύω, μειώνω το αποτύπωμα του άνθρακα, μειώνω τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και όπως σας είπα τα χρήματα τα οποία θα εξοικονομήσω μπορεί να χρησιμοποιηθούν για κάτι άλλο. Αυτή λοιπόν είναι η υποτιθή η θετική προστιθέμενη αξία για την επιπλέον μόνωση σε κτίρια ή τη θερμομόνωση των κτίριων. Ε, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να συνεισφέρουμε στη στρατηγική Ευρώπη 2020. Κάτι επιπλέον. Πολλές φορές ένα σχολείο θα πρέπει να αποφασίσει αν ε, θα χρησιμοποιήσει τα κονδύλια τα οποία διαθέτει για ευφυή παιδεία ή για ε, καλύτερη θερμομόνωση του κτηρίου. Η θερμομόνωση είναι μια επένδυση και η οποία θα μου εξοικονομήσει χρήματα διότι θα έχω εξοικονόμηση ενέργειας και επομένως μπορώ να επενδύσω τα χρήματα αυτά στη συνέχεια για ευφυή παιδεία. Ευχαριστώ. Thank you ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να σταθώ σε ένα μόνο στοιχείο του εγγράφου σας και σας το παραθέτω λέει οι τοπικές περιφερειακές και δημόσιες αρχές θα πρέπει να είναι εταίροι ε, και ενδιαφερόμενοι. Έγγραφο από τον Απρίλιο του 2012 CMR, e του CMR. Εκεί λέτε ότι είναι οι απόψεις του CMR για την υποστήριξη της εδαφικής συνοχής. Και αναφέρεστε στην υφιστάμενη κατάσταση για την πιθανή χρηματοδότηση για τη συνοχή. Και έχετε ένα σημείο 1 που λέτε ότι χαιρόμαστε ότι ε, έχει ληφθεί υπόψη ε, και έχει παραμείνει ο στόχος για την εδαφική συνοχή. Τέλος παράθεσης. Και αυτό φυσικά ισχύει μόνο εν μέρη, διότι αν ε, υπολογίσουμε την πρόταση συνοχής που έγινε το καλοκαίρι πέρσι, και τα κονδύλια για τη συνοχή, ε, αποκλείοντας το Connecting Europe. Είναι δύσκολο βέβαια να πούμε αν θα πρέπει να το ή να το αποκλείσουμε. Τα κονδύλια αυτά ε, σε σχέση με το παρελθόν είναι μείον 5,1%. Και γι' αυτό και στο δεύτερο τμήμα του κειμένου σας αναφέρεστε σε απορρόφηση των ε, κονδυλίων στα σημεία 7, 8 και 9, είστε πολύ αρνητικοί ως μέλη του CMR για την ε, απορρόφηση κατά να Έχετε ένα ποσοστό 2,5 του ΑΕΠ και λέτε ότι δεν αντικατοπτρίζει την κατάσταση. Δύο πράγματα. Αυτό το 2,5% προκύπτει από αυτά τα λιγότερα κονδύλια. Θα είναι θαύμα να δοθούν περισσότερα κονδύλια, δεν νομίζω ότι θα δοθεί. Ε, ε, το 2,5% πολύ είναι πραγματικά. Και παρόλο που επί της αρχής υποστηρίζω τις προτάσεις σας για αυτό το 2,5%, το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι τα κονδύλια δεν θα είναι σε καμία περίπτωση τα ίδια με αυτά που έχουμε αυτή τη στιγμή, διότι η κατάσταση πόρο απέχει από το να χαρακτηριστεί εύκολη, έχουμε κρίση και δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να έχουμε ε, ανοιχτό το περιθώριο. Εδώ έχουμε από το 3,2 στο 3,7 ανάλογα με το πόσο καλή είναι η επίδοσή σας. Αν είστε στο 75 παίρνετε 3,2. Αν είστε στο λιγότερο παίρνετε 3,7. Αν εφαρμόσετε λοιπόν την αρχή που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν ξέρω αν θα την αλλάξουν, μπορεί και να μην την αλλάξουν. Ε, δεν έχει καμία σχέση όμως αυτός με τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές, διότι από το 2,5 με 0,5 από τις δύο πλευρές θα είναι από το 2,25 μέχρι το 2,75 δεν θα ξοδεύουμε ή θα δαπανούμε ή ξεκονομούμε περισσότερα χρήματα, αλλά προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη τουλάχιστον αυτά που γράφετε στα 8 σημεία σας. Ε, ότι υπάρχουν ακόμα πολύ μεγάλες διαφορές για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές ε, και θα πρέπει να λάβουμε και αυτές υπόψη. Ε, και αυτή είναι η πρότασή μου, θα πρέπει να το σκεφτείτε, διότι το να ζητάτε υψηλότερο το ανώτατο όριο δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε να το επιτέχουμε. Υποστηρίζω τους εισηγητές, την κυρία Κρέλ ε, και τον κύριο Φανίστερ ε, αλλά αν κάτσουμε να καταγράψουμε τον κατάλογο των πόλεων, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο θα είναι ε, και, το πολιτικό κόστος. Κανένας δεν ξέρει πώς έχει κατάσταση ε, και πώς αλλάξει στην κάθε χώρα. Όλα αυτά έχουν μια δυναμική, αλλάζουν συνεχώς και ε, αν ε, αλλάξουν και οι ισορροπίες στις περιφέρειες καταλαβαίνετε πόσο δύσκολα θα τα πράγματα το αλλάξουμε σε νέους φορείς που μπορεί να αλλάξουν, ε, τότε μπορεί να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά αν καταγράψουμε κατάλογο των πόλεων, τότε θα πρέπει να εφαρμόσουμε διαφορετικά κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να καθοριστούν ακριβώς αυτό τον κατάλογο των πόλεων. Γι' αυτό ακριβώς ε, διαφορώ ε, με αυτό που είπατε εσείς και θα υποστηρίξω τους εισηγητές μας σε αυτή την περίπτωση. Ευχαριστώ πολύ. Yeah, uh, thank you, ευχαριστώ. Συμφωνώ βεβαίω και υποστηρίζω τι προτάσει και τι ιδέε που προτείνουν οι συνάδελφοι από τις διαφορέ περιφερειακέ, οργανώσεις τις οποίες επίσης υποστηρίζω στους στόχους τους. Θα ήθελα ωστόσο να διατυπώσω την ίδια κοινή ερώτηση προς όλες τις παρουσιάσεις. Πώς θα επιτύχουμε τους στόχους αυτούς. Μιλήσατε παραδείγματι για το ρόλο των περιφερειών που πρέπει να είναι πολύ σημαντικός. Η κυρία Ζαμπάρη είπε παραδείγματι ότι οι θεματικές ιδέες θα πρέπει να προσδιορίζονται σε περιφερειακό επίπεδο και συμφωνώ βεβαίως. Ρωτάω όμως τους συναδέλφους πώς θα το επιτύχουμε. Ασφαλώ η Επιτροπή μα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα προσπαθήσει να υπογραμμίσει, να ενισχύσει δηλαδή, τη διατύπωση ε, στο κείμενο ε, αλλά πρέπει να ξεπεράσουμε τις λέξεις και να περάσουμε σε δράση, δηλαδή σε ουσιαστική επίτευξη αυτού του στόχου. Γι' αυτό θα ήθελα να μου δώσετε κάποιες ιδέες. Και για τον κύριο Τσίλσλι. ο οποίο είναι, αν κατάλαβα καλά, κύριε Τίλσλι, είστε αναπληρωτή από τι εκλογέ τη προηγούμενη εβδομάδα. Α, αν, αν κερδίσατε, δεν σα συγχαίρω πάντω. Σκόπευα σα συγχαρώ, αλλά δεν σα συγχαίρω. Εν πάση περιπτώσει είναι σημαντική οικονομική ε, παράγοντες στα αστικά κέντρα και πρέπει να υποστηριχθούν. Οι επενδύσει, ωστόσο, στα αστικά κέντρα, στι αστικές περιοχές δεν θα πρέπει να αποβαίνουν μόνο όφερος στις ίδια της πόλης. Θα πρέπει να ε, βοηθούν ολόκληρη την περιοχή γύρω από αυτήν. όπω θέλετε πείτε την, είτε είναι λειτουργικό αστικό κέντρο, είτε είναι ακόμα και ύπεθρος γύρω από το κέντρο, από το αστικό κέντρο, πρέπει να αποβαίνει όφελος του αυτή η βοήθεια. Και ρωτώ τον κύριο Τίλτσλι πώ μπορεί να το εξασφαλίσουμε αυτό, πώ μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα επωφεληθούν μόνο από τι επενδύσει αυτέ τα αστικά κέντρα και επίσης ε, στην ιδέα για ένα κατάλογο, ένα κατάστοιχο πόλεων θα ήθελα να πω ότι δεν συμφωνώ και εγώ όπως και οι άλλοι συνάδελφοι. Εμείς στην Ουαλία από την οποία κατάγομαι δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα ως προς την ε, κατάρτιση του καταλόγου γιατί είναι μικρά τα αστικά μας κέντρα αλλά νομίζω θα ήταν πολύ καλύτερο να εξασφαλιστεί ε, μια δυνατότητα συμμετοχής για τα αστικά κέντρα ώστε αυτά να μπορούν να προσδιορίσουν και να ορίσουν το μέλλον τους. Ευχαριστώ. Αλφονσί. Ευχαριστώ. Δύο παρατηρήσεις έχω να κάνω. Σε ό,τι αφορά τη μακροαιρεσιμότητα καταρχήν, ξέρετε ότι συμφωνούμε με τις επικρίσεις κατά της πολιτικής αυτής και της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Λετριάνο είπε ότι η Γαλλία είναι ένθερμη υπέρμαχος αυτής της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας, αλλά οι πολιτικές συνθήκε έχουν αλλάξει φαίνεται οριστικά. Οπότε μήπως ε, τροποποιηθεί και η σχέση της Γαλλίας ω προς αυτό. Άλλο θέμα, Εταιρικέ σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, κρατών και τοπικών και περιφερειακών αρχών. Φυσικά βασικός εταίρο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που καθορίζει προτεραιότητες και οι περιφέρειες θα καθορίσουν τις ανάγκε του, θα προσδιορίσουν ανάγκε του και μεταξύ του διαλόγου μεταξύ προτεραιτήτων και αναγκών των περιφερειών θα έχουμε καλά λειτουργικά προγράμματα και αγαστά αποτελέσματα για την πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης. Ε, βέβαια, φαίνεται ότι δίνουμε υπερβολική έμφαση σε αυτές τις εταιρικές σχέσεις, συμβάσεις σχέσεις και ελπίζω με τη βοήθεια των εισηγητών ε, να έχουμε όσο δυνατόν περισσότερη ανάμειξη των περιοχών, των περιφερειών σε αυτές τις συμβάσεις εταιρικής σχέσης και να δούμε πώς θα καταφέρουμε να έχουμε άμεση διαπραγμάτευση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και, και περιφερειών, χωρί να περνάμε από την κεντρική διοίκηση. Γιατί στα πλαίσια του πολιτού χρηματοπιστωτικού πλαισίου, του δημοσιονομικού πλαισίου που καθυστερημένα προσδιορίζουμε λόγω των οικονομικών ε, δυσχεριών, ε, θα έχουμε πολύ λίγο χρόνο για τις διαπραγματεύσεις, γιατί το 2013 θα έρθει αμέσω ε, και δεν θα πρέπει σε αυτόν τον περιορισμένο χρόνο να, να σπεύσουμε και από υπερβολική ταχύτητα να κάνουμε λάθη που θα μας βαρύνουν μετά σε όλη την επόμενη ε, περίοδο δημοσιονομικών προοπτικών. Προσοχή λοιπόν σε αυτό το μηχανισμό για να έχουμε πραγματικά λειτουργικά προγράμματα. Τέλος, σε ό,τι αφορά την ανάγκη διάκρισης μεταξύ των προσεγγίσεων ανάλογα με τι ιδιαιτερότητε των περιοχών. Γιατί υπάρχουν μεγάλε ανισότητε και διαφορέ. Πάντω, το μοναδικό κριτήριο που λαμβάνεται υπόψη φαίνεται ότι είναι το αναπτυξιακό κριτήριο. Ενώ υπάρχουν και άλλε ιδιαιτερότητε που είναι πολύ ισχυρέ. Για παράδειγμα, η θέση Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν δείχνει κανένα ενδιαφέρον για την ε, εφαρμογή του άρθρου 174 για τις ε, ιδιάζουσες περιοχές, όπως ε, τις νησιώτικες, και το λέω γιατί και εγώ κατάγομαι από τέτοια περιοχή, νομίζω θα μπορούσε να είναι πολύ πιο πρωτότυπη και φάνταστη στην πρόταση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ό,τι φορά το αποθεματικό επίδοσης που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα περιφερειακά προγράμματα. Αν στόχος σας είναι μια πλειοδότηση υπέρ της παραγωγικότητας δεν είναι και πολύ ενδιαφέρον. Αν θέλετε όμως πραγματικά να λάβετε υπόψη το ρυθμό προσαρμογής και τι ιδιαιτερότητες των ε, περιφερειών ε, θα πρέπει να το εξετάσουμε. Άρα να δούμε πώς θα προσαρμοστεί τέτοια πρόταση αποθεματικού επίδοσης για τις άκρος ιδιάζουσες περιοχές. Ε, προσοχή λοιπόν γιατί μια μια όμορφη πολιτική για 500 εκατομμύρια απόλυτο δεν θα είναι σωστή. Ο κύριος Βλάσακ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας δώσατε να εξετάσουμε όλα αυτά τα πολύ σημαντικά ζητήματα με εκπροσώπους των περιφερειακών ενώσεων και οργανώσεων. Και θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω θερμά τους συνεισηγητές μας που έλαβαν υπόψη τα σχόλια των προσκεκλημένων μας και έχω και κάποιες ερωτήσεις. Πώς αξιολογείται την αρχή της εταιρικότητας, πώς περιλαμβάνεται η αρχή αυτή στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είστε ικανοποιημένοι, θεωρείτε επαρκή αυτή την πρόταση για την εταιρικότητα. Δεύτερον, δεν έχετε την αίσθηση ότι δεν υπάρχει δέους αντιπροσωπευτικότητα των περιφερειών σε ό,τι αφορά την επικοινωνία τους με τα κοινοτικά θεσμικά όργανα, το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απροκειμένου. προκειμένου. Και τρίτη ερώτηση για τα πιθανά εμπόδια που θα υπάρξουν στις ε, συμβάσεις εταιρική σχέσης. Νομίζω ότι στην περίπτωση αυτή μπορούμε να αξιοποιήσουμε το, την τεχνική αρρωγή σε επίπεδο κρατών μελών. Νομίζω ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή την τεχνογνωσία. Ποια είναι η γνώμη σας. Ευχαριστώ. Thank you very much. At this point, I'd like to give the floor. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον πρόεδρο της ε, Επιτροπής ε, Περιφερειακών Υποθέσεων του της Τοπικής Βουλής της Τοσκάνης, τον κύριο Ταραντάς. Δύο-τρία λεπτά παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόμως της Αρχής Διαχείρισης της περιοχής της Τοσκάνης, ε, λαμβάνω το λόγο ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του ε, Περιφερειακού Συμβουλίου της Τοσκάνης και θέτω τρία ερωτήματα που αφορούν τη μακροοικονομική ερωσιμότητα, τις εταιρικέ σχέσεις και τις συμβάσει τους και το σύστημα χρηματοοικονομικής διαχείρισης. Πρέπει να σας πω ότι είμαστε σύμφωνοι με πολλέ από τι εκτιμήσεις που ακούστηκαν και από τους συζητητέ, αλλά και από πολλούς από τους προλαλήσαντες. Για τη μακροοικονομική ερεσιμότητα, η περιοχή της Τοσκάνης θεωρεί ότι το να δεσμεύσουμε την πολιτική συνοχή βάση μακροοικονομικών στόχων που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση για την Οικονομία στην ε, σε εθνικό επίπεδο αντιβαίνει ε, με τους οικονομικούς όρους, διότι οι πόροι της ανάπτυξης και των θέσεων αποσχόλησης δεν μπορεί να δεσμεύονται και να καθορίζονται από την οικονομική και νομισματική σταθερότητα. Πρέπει να γίνει διάκριση λοιπόν μεταξύ της πειθαρχίας που είναι απαραίτητη, που ε, είναι απαραίτητη από πλευράς περιφερειών και από ένα μπλοκ που μπορεί να δοθεί μακροοικονομικά και που αποτελεί πρόσκομα για την ανάπτυξη. Βιώνουμε αυτή τη στιγμή μια οικονομική οικονομική χρήση που ελοχεύει ο κίνδυνος να γίνει και πολιτική κρίση και γι' αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε ε, με, από τα σπάργανα να σκεφτούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση γεννήθηκε ως μία ομοσπονδιακή ένωση και θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη ότι δεν μπορούμε να λαμβάνουμε μέτρα τα οποία μπορεί να αντιβαίνουν την ε, δημοκρατία. Εμείς υποστηρίζουμε λοιπόν το άρθρο 44 στο σχέδιο των ε, εισηγητών. Δεύτερον, για τι συμβάσει εταιρική σχέση. Το άρθρο 5 είναι το βασικό ε, άρθρο που αναφέρεται στα διαρθρωτικά ταμεία και προασπίζει και τα δικαιώματα των περιφερειών. Αλλά ξέρουμε ότι στο Συμβούλιο υπάρχουν κάποιοι προσανατολισμοί να μειωθεί η βαρύτητα αυτού του άρθρου και ουσιαστικά να αποκλείσουμε ε, ή τουλάχιστον να είναι λιγότερη η συμμετοχή των ε, τοπικών και περιφερειακών αρχών στις ε, βάσεις εταιρική σχέσης. Ακούστηκε από πολλούς, ενώ εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να προασπίσουμε την κοινή μάλιστα πλήρως των περιφερειών και συμφωνούμε με τις τροπολογίες που παρουσίασαν οι συγητές προς αυτή την κατεύθυνση. Τέλος, το οικονομικό σύστημα, το χρηματοοικονομικό σύστημα. Εδώ είναι πιο περίπλοκα και πιο τεχνικά τα θέματα, αλλά εμείς θεωρούμε ότι το θέμα της διαχείρισης, ε, όπως και το θέμα της κοινή αγροτικής πολιτικής ε, και της διαχείρισης ε, για τα διαρθρωτικά ταμεία είναι λανθασμένη κίνηση, διότι οι παρεμβάσεις είναι διαφορετικές και οι ενισχύσεις δεν είναι συμβατές. Για τα διαρθρωτικά ταμεία θα πρέπει οι επιδοτήσεις να λαμβάνονται υπόψη βάσει και της ε, διάρκειας και δεν μπορούν να γίνονται οι αιτήσιες ε, διορθώσεις και οι έλεγχοι που γίνονται στη γεωργική πολιτική. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ε, minutes for the commission, please. Ευχαριστώ και δύο-τρία λεπτά στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Θα ήθελα εκ μέρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να ευχαριστήσω την Επιτροπή ΡΕΚΙ για την διοργάνωση αυτή τη συζήτηση. Είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε τις απόψεις των εκπροσώπων των περιφερειακών οργανώσεων και έχω την αίσθηση ότι η προτάσει Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν πολύ καλό σημείο αφετηρίας και έτυχαν αρκετά μεγάλη υποστήριξη. Άλλωστε, στόχο τη συζήτηση είναι να βελτιωθούν ακριβώ αυτέ οι προτάσει. Και από αυτή την άποψη με ιδιαίτερη χαρά ακούσαμε τις παρεμβάσεις των προσκεκλημένων και των μελών της Επιτροπής. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα ζήτημα που είναι κεντρικό. Διανύουμε πολύ χαλεπούς καιρούς οικονομικά και γνώμη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι η πολιτική συνοχή θα διαδραματίσει θεμελιώδη ρόλο για να ε, ενισχύσουμε την οικονομική ανάπτυξη και να δημιουργήσουμε θέσει απασχόληση. Χρειαζόμαστε όμω δύο συνιστώσει για να το επιτύχουμε αυτό. Η πρώτη συνιστώσα, το πιο πρώτο συστατικό, είναι συσχετισμό με την στρατηγική του 2020 ε, στοχοθέτηση των πόρων και στενή συνεργασία σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Τα χρειαζόμαστε από κοινού και τα δύο. Χρειαζόμαστε και τι δύο συνιστώσει. Δεν μπορούμε να έχουμε συγκέντρωση χωρί περιφερειακή ανάπτυξη, ούτε μπορούμε να έχουμε περιφερειακή ανάπτυξη χωρί προηγούμενη συγκέντρωση των προτεραιοτήτων. Οπότε. Ερχόμαστε στα θέματα των συμβάσεων εταιρική σχέση και πώς θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και εμπράκτος. Θα ήθελα να επαναλάβω κάποια σχόλια που ακούσαμε. Κατά τη γνώμη μα, η συμβάση εταιρική σχέση δεν είναι εταιρική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, κράτου μέλου, αλλά μια συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, κράτους μέλους, ε, εκ μέρου των εταίρων όμως που θα είναι, δικαιού, που θα είναι οι συμβαλόμενοι αυτής της συμφωνίας. Ο κύριος Ζέλερ ρώτησε πώς θα εξασφαλίσουμε την εφαρμογή της εταιρικότητας μέσω του άρθρου 5 που προβλέπει νομική υποχρέωση της ε, θέσπης αυτής της εταιρικότητας. Και φυσικά θα είμαστε πολύ προσεκτικοί στη δίρυση των ενωμών υποχρεώσεων, στη συζητήση με τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή των προγραμμάτων. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ερώτηση του κυρίου Αλφόνση για την ανάμειξη των περιφερειών και το με ποιο τρόπο θα γίνουν. Η συμβάση εταιρική σχέση είναι ένα μηχανισμό μεταξύ άλλων μηχανισμών. Και η διαπραγμάτευση των επιχειρησιακών προγραμμάτων εναπόκειται στη διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών. Και τα κράτη-μέλη που έχουν ισχυρή περιφερειακή δομή ε, θα διεξαγάγουν αυτές τις διαπραγματεύσεις και μερικές φορές οι διαχειριστικές αρχές σε εθνικό επίπεδο είναι περιφέρειες, οπότε είναι πολύ σημαντικός ο διαχειριστικός ρόλος τους στα διάφορα αυτά επιχειρησιακά προγράμματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη θεματική συγκέντρωση. Φυσικά, η θεματική συγκέντρωση θα πρέπει να λάβει υπόψη τις ε, διαφορές, τις ιδιαίτερες ανάγκες των περιοχών, Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε εθνικό επίπεδο, κατηγορία περιφερειών. Οπότε κάθε κράτος έχει περιθώριο λιγμών ε, προσαρμόσει την θεματική συγκέντρωση στις ε, μεμονωμένες ε, ανάγκες και ιδιαιτερότητες των περιφερειών του. Σε ό,τι αφορά τώρα τη μακροοικονομική αιρεσιμότητα, σχετικά καθόδε ζήτημα, θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν αφορά μόνο την εμπλοκή των κονδυλίων ή την πάυση της ροής των κονδυλίων. Είναι ένας προοδευτικός σταδιακός μηχανισμός που στόχο έχει να δημιουργήσει διασυνδέσεις μεταξύ διαφορετικών οικονομικών θεμάτων. Στο άρθρο 21 προβλέπεται το πρώτο στάδιο που είναι ο διάλογος μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κράτους μέλους για τις συμβάσει εταιρική σχέση. Και μια και θεωρούμε ότι η συμβάση εταιρική σχέση είναι ένα μηχανισμό που εμπλέκει τα κράτη-μέλη διαφορε φορέ και τι ε, ε, περιφέρειε, τότε βλέπουμε ότι είναι περίπλοκη διαδικασία. Το θέμα των κυρώσεων και των διακοπών, των αναστολών είναι ένα ζήτημα που θα εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε έσχατο βαθμό μόνο, ω έσχατη λύση. Και επανέρχομαι στο θέμα τη πλατφόρμα ε, ανάπτυξη των πόλεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρότεινε μια τέτοια πλατφόρμα ανάπτυξη των πόλεων, γιατί ε, θεωρούμε ότι έχουμε αρκετά θεσμικά όργανα, αρκετές οργανώσεις, δεν χρειαζόμαστε ένα νέο ε, θεσμό. Αλλά διαπιστώσαμε ανάγκη ενίσχυση του δυναμικού προαγωγής της ανταλλαγής ε, εμπειριών, όπως είπε και ο κύριος Τίλση, μεταξύ των φορέων της αηφόρων ανάπτυξη των πόλεων ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των προγραμμάτων. Θεωρούμε ότι υπάρχει τέτοια ανάγκη Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστώ. Thank you very much indeed. Σας ευχαριστώ θερμά. Και τώρα συνεχίζουμε ως εξή. Δίνουμε τον λόγο σε όλους τους προέδρους, σε όλους τους παρόντες και αν έχουμε χρόνο θα ακούσουμε και τους συναδέλφους και πάλι. Ο κύριος Λεντιχιάν παρακαλώ. Πρόεδρε, σα ευχαριστώ θερμά. Ε, θα ήθελα ξεκινώντα να ευχαριστήσω όλους όσοι έλαβαν το λόγο για την ε, συμμετοχή τους στη συζήτηση και πάνω απ' όλα βέβαια για τη ε, σημεία σύγκληση τα οποία σημειώθηκαν κατά τη συζήτηση. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι εδώ βρίσκομαι ως Πρόεδρος της διάσκεψη των απομακρυσμένων και θαλάσσιων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν εκπροσωπώ ούτε την τρέχουσα ούτε τη μελλοντική κυβέρνηση της Γαλλίας και τη βέβαια έχω τις δικές μου πεπιθήσεις. Θα ήθελα να πω ότι για τις περιφερειακές απομακρυσμένες και ε, άκρως απομακρυσμένες περιφέρειες Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήθελα να πω ότι τις προτάσεις τις οποίες διατυπώνουμε, τις διατυπώνουμε ακριβώς επειδή εκπροσωπούμε από απομεμακρυσμένες και θαλάσσιες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μια παρατήρηση που ακούσαμε και από τον εκπρόσωπο της Ουαλίας ή των ορεινών περιοχών. Έχουμε ανησυχίες με λύματα κοινά να εκφράσουμε στο σύνολο των απομακρυσμένων και θαλασσίων περιφερειών. Γι' αυτό προτείνουμε τη σχετική τροπολογία που αφορά τα νησιά και γι' αυτό εκφράζουμε την ανησυχία μας ως προς το σύστημα των υποδομών, την αναγνωσιμότητα των ε, ε, υποδομών για όλες τις περιφέρειες, μάλλον την αιρεσιμότητα των, υποδομών για όλες τις περιφέρειες, είτε είναι πιο πλούσιες είτε λιγότερο ευμαρείς, ακριβώς για να έχουν την ίδια δυνατότητα πρόσβαση στην ε, ανάπτυξη. γιατί θα έλεγα ότι με ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα στο ίντερνετ υψηλής ταχύτητας, εάν μια περιφέρεια είναι πλούσια ούσα απομεμακρυσμένη είναι σε μειονεκτική θέση σε σχέση με την εισαγωγή του ε, ταχαίου ε, ίντερνετ, του υψηλής ταχύτητας ίντερνετ. Αλλά αυτό δεν ισχύει μόνο για το ίντερνετ, αλλά γενικότερα για τις μεταφορές. Και αυτό θα ήθελα να το υπογραμμίσω ως στόχο της οργάνωσης των απομακρυσμένων και θαλάσσιων περιφερειών. Επίσης, Μας ενδιαφέρει η θεματική οργάνωση, η θεματική συγκέντρωση Ίσως κάποιο θεωρούσε ότι εμεί προσπαθούμε να κατακαιρματίσουμε, ότι προτιμούμε τον κατακαιρματισμό τη θεματολογία ως οργάνωση. Όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό. Θέλουμε να είναι ολοκληρωμένη, ενοποιημένη η θεματολογία, αλλά αρκετά ανοιχτή, ώστε να επιτρέπει και την εξειδίκευση, την ιδιαιτερότητα για την κάθε περιφέρεια, με στόχου την ενέργεια, την έρευνα και την Ευρώπη βέβαια 2020. Εγώ δεν βλέπω σε αυτό καμιά απόκληση μεταξύ αυτών των, τα οποία είπα εγώ και των όσων άκουσα από τους λοιπούς ομιλήσαντες για την συγκέντρωση θεματολογική. Απλώς υπογράψω ότι πρέπει να είναι ευφυής αυτή η συγκέντρωση. Ιδάλλως δεν θα έχουμε κάποιον συνομιλητή από την άλλη πλευρά για να συζητήσουμε τι σημαίνει αυτό σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, στο θέμα της εταιρική σχέσης και ιδιαίτερα της Παρατηρήσει και ερωτήσει κυρίω του κ. Ολμπρίχτ στο ίδιο θέμα, αλλά και κάποιων άλλων βουλευτών. Θα ήθελα να πω ότι για μα, για τη διάσκεψη των απομακρυσμένων και θαλάσσιων περιφερειών, πρέπει ο κώδικα συμπεριφορά να είναι ευρωπαϊκό. Είχε αρχικά συμπεριληφθεί, μετά βγήκε από την πρόταση. Θα θέλαμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τον επαναφέρει στο τελικό κείμενο. Ιδάλω, ο κίνδυνος να παραμεληθεί η περιφερειακή διάσταση και ταυτότητα στην εταιρική σχέση είναι πολύ υψηλό. Θέλουμε λοιπόν ο κώδικας συμπεριφοράς να σωματωθεί στον κανονισμό και να είναι ευρωπαϊκός. Τουναντίον για την εύρυθμη λειτουργία τη εταιρική σχέσης ε, η διάσκεψη των απομακρυσμένων και θελάσσιων περιφερειών τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ιδιαίτερα υπογραμμίζει προτάσεις της την έννοια της εδαφικής εταιρική σχέσης, που σημαίνει ότι πέραν της εταιρική σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών για τη νέα γενεά ταμείων, ταμείων συνοχής, θα πρέπει να υπάρχει ένα εδαφικό σύμφωνο μέσα σε κάθε κράτος μέλος, ανάλογα με την ιδιαιτερότητά του κράτους, ανάλογα με τον αριθμό των περιφερειών του κτλ. Ένα σύμφωνο όμως εδαφικό για το κράτος μέλος, το οποίο θα προσφέρει μια μορφή εταιρικής σχέσης για ουσιαστική, λειτουργική και όχι απλώς τυπική επικουρικότητα. Και επίσης για την μακροοικονομική ρεσιμότητα θα ήθελα να πω ότι η ΔΑΘΠΟ διάσκεψη απομακρυσμένων και θαλάσσιων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι επί της ουσίας υπέρ της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας, αλλά ξέροντας ότι αναγκαστικά θα πρέπει να προβούμε σε συμβασμούς, προτείνουμε συμβαστικά αυτή την πρόταση για να διαφυλάξουμε και τα συμφέροντα των περιφερειών που εκπροσωπούμε στη διάσκεψή μας, με βάση και τα όσα σας είπα εισαγωγικά και τις τροπολογίες βεβαίως που εξέθεσα. Αυτά πιστεύω ότι ήταν τα κύρια ζητήματα στα οποία έπρεπε να δώσω απαντήσεις ε, στις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ πάντως που μας παρακολουθήσατε, που μας ακούσατε και ελπίζω ότι θα λάβετε υπόψη στο μέλλον και τις ανησυχίες των απομεμακρυσμένων και θαλάσσιων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις στα θέματα της πολιτικής συνοχής. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ε, παρουσίαση, την απάντηση στα σχόλιά σας. Η κυρία Μισελ Σαμπάν παρακαλώ τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ μετά τον κύριο Λιτριόν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και όλες για τις ερωτήσεις και ενδεχομένω τις παρατηρήσεις που μας διατυπώσατε σε αυτή τη συζήτηση. Διαπίστωση είναι βεβαίως ότι υπάρχει αίτημα, υπάρχει προσδοκία από πλευράς των περιφερειών να δοθούν απαντήσεις όλα αυτά ερωτηματικά, να ακουστεί η πρότασή τους για όλα αυτά τα ζητήματα. Γιατί βεβαίω ο ρόλος τους είναι καθόριστικη σημασία και θα είναι και στους επόμενου μήνε και χρόνια. Θα ήθελα εγώ ιδιαίτερα να παρέμβω σε ένα-δύο σημεία. Γιατί συμφωνώ σε πολλά με τον κύριο Λιθιό. Να επικεντρωθώ όμω εγώ στην θεματολογική συγκέντρωση την οποία υποστηρίζουμε, που όμως θα πρέπει τότε να επιτρέπεται η αναγνώριση των εδαφικών ιδιαιτεροτήτων ε, με τρόπο ευφύ για να, για μην, για να μην γίνει αυτός ο κατακαιρματισμός, για να μην χαθεί η ιδιαιτερότητα δηλαδή, των περιφερειών μας, θα πρέπει να ε, υπάρχει αυτή η θεματολογική συγκέντρωση για να αποφευθεί και ο κατακαιρματισμός βεβαίως των κονδυλίων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις περιφέρειες, για την Ένωση, για τη Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης που εκπροσωπώ και που υποστηρίζει τις, ε, τα συμφέροντα των περιφερειών, γιατί βεβαίω τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικά συμφέροντα από τις περιφέρειες. Ξέρετε ότι έχουμε περιφέρειες σε διαφορετικά επίπεδα αρμοδιοτήτων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση με διαφορετικές αρμοδιότητες και νομοθετικές. Μερικές φορές δηλαδή είναι μικροκράτη οι περιφερειές μας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις δεν έχουν τέτοιες αρμοδιότητες περιφέρειες και άρα πρέπει αυτήν την ιδιαιτερότητα να τη λαμβάνουμε υπόψη μας προς την εταιρική σχέση. ερώτημα προς μια κοινή ε, πρόταση και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τεχνική στήριξη βεβαίως, δεν έχουμε καμιά αντίρρηση, την υποστηρίζουμε γιατί θα μας επιτρέψει και να διευρύνουμε το πεδίο των ε, δραστηριοτήτων μας και να γνωστοποιήσουμε περισσότερο το σύνολο, στο σύνολό τους τις αρμοδιότητες των ε, περιφερειών. Κλείνοντα, θα ήθελα να πω ότι πιστεύουμε πω θα δοθεί ευκαιρία και για άλλε συνεδριάσει, για άλλε συναντήσει και επαφέ για να επεξεργαστούμε τις προτάσεις αυτές στη συνέλευση των περιφερειών της Ευρώπης θα ήθελα να υπενθυμίσει και είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε να κάνουμε με περιφερειακή πολιτική. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με περιφέρειες που συνεργάζονται με περιφέρειες και συνεργάζονται μέσα στις περιφέρειες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να δει και ο πολίτης πώς αρχή αυτή της ε, επικουρικότητας την οποία προσπιζόμαστε μπορεί ουσιαστικά να λειτουργήσει και να υλοποιηθεί. Και για να κλείσω θα ήθελα να πω ότι από πλευρά μα, από πλευρά τη ε, Συνέλευσης των Περιφερειών είμαστε υπέρ τη διαφύλαξη και ανάπτυξη μια αποτελεσματική εταιρική σχέση με την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για τα σχόλιά σας. Και τώρα η κυρία Γκόνορσον έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους για τα πολύ ενδιαφέροντα σχόλια που ακούστηκαν. Θα σχολιάσω τρία διαφορετικά πράγματα από τα όσα ακούστηκαν και τις ερωτήσεις που μετέθησαν. Καταρχάς, τη σχέση μεταξύ κράτους και περιφερειών. Ε, ανησυχώ λίγο για κάποια από τα πράγματα που ακούω. Ακούμε τις μεγάλες πόλεις και λέμε ότι οι μεγάλες πόλεις είναι ο κινητήριος μοχλός της ανάπτυξης. Εμείς στην νομοθεσία μας θα πρέπει να επικεντρωθούμε ε, στην ε, σχέση μεταξύ κράτους και περιφερειών και θα πρέπει... Ε, να δούμε και τη σημασία των τοπικών αρχών ε, για θέματα διάθεσης απορριμμάτων, ε, ενεργειακά ζητήματα περιβαλλοντικά, εφοδιασμού τροφίμων, ε, ε, της φύσης, της ψυχαγωγίας και θα πρέπει επίσης να γνωρίζουμε ότι η ανάπτυξη αυτή τη στιγμή δεν συμβαίνει απλώς και μόνο στις μεγάλες πόλεις. Σε πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το μεγαλύτερο τμήμα της ανάπτυξης του ΑΕΠ προκύπτει από τις μικρότερες πόλεις, ε, τα χωριά και τις περιοχές της υπαίθρου. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πώς οι πόλεις και οι περιοχές της υπαίθρου μπορούν να συντεριαστούν ε, στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής. Και θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο και τη χρησιμότητα του στρατηγικού πλαισίου διότι μέσω καλύτερου συντονισμού των διαφόρων ταμείων θα μπορέσουμε να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα και φυσικά πολύ καλύτερη χρήση των πόρων που επενδύονται και των όσων κάνουμε. Και είναι αυτός τελείως διαφορετικός τρόπος ε, να εξετάσουμε την εδαφική συνοχή. Ε, έχουμε μια προσέγγιση προς τα πάνω και δεν τα βλέπουμε όλα κατακαιρματισμένα. Θεωρούμε ότι ε, θα πρέπει λοιπόν ε, για τα θέματα της εδαφικής συνοχής να έχουμε νομοθετική πράξη επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην εκχωρείται αυτή η αρμοδιότητα στα κράτη-μέλη. Τέλος, για την εταιρική σχέση, θεωρούμε, όπως σας είπα και πριν, ότι χρειαζόμαστε έναν ευρωπαϊκό ορισμό της εταιρική σχέσης και αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνεται στον κώδικα δεοντολογίας. Γνωρίζουμε ότι από πλευράς κρατών μελών ερίζουν οι απόψεις για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να λειτουργούν αυτές οι εταιρικέ σχέσεις, ερίζουν οι απόψεις για τον τρόπο με τον οποίο ε, θα πρέπει να συμπεριληφθούν και το τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο ως εταίροι και όχι ως ομάδες ενδιαφερόντων και ομάδες συμφερόντων. Ε, γι' αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε ένα σαφή ορισμό του τι ακριβώς είναι εταιρική σχέση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πολ Τίσλι τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ακούστηκαν τόσα πολλά σχόλια που πραγματικά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να απαντήσω στα περισσότερα από αυτά. Θα κάνω όμως μία απόπειρα να απαντήσω σε δύο πτυχές. Την ευφυή εξειδίκευση και τον ε, κατάλογο αυτών ε, των πόλεων. θεωρούμε ότι τα προγράμματα θα μπορέσουν να εντοπίσουν ποιες είναι ε, οι αδυναμίες αλλά και ποια είναι και τα μοναδικά χαρακτηριστικά που έχει κάθε περιοχή και κάθε περιφέρεια. Η εφηβής ε, εξειδίκευση είναι ακριβώς τμήμα μιας τέτοιας στρατηγικής και θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική στις μητροπολιτικές περιοχές. Η ανάπτυξη των αστικών περιοχών βάσει μια συγκεκριμένη βάση ε, γνώσεων και τομεακή ανάπτυξη ε, και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα αυτά ε, για την εξέλιξή του. Οι πόλει θα πρέπει λοιπόν να διαθέτουν μέσα όπω είναι το ITI για να αναπτύξουν κατάλληλα προγράμματα τα οποία θα μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα χώρο στον οποίο θα μπορέσουμε να έχουμε αποτελεσματικές εταιρικέ σχέσεις και με πανεπιστήμια αλλά και με μεγάλες επιχειρήσεις και εργοδότες ώστε να έχουμε πιο αποτελεσματικά στοιχεία και ολοκληρωμένες δραστηριότητες, ιδίω αυτές που υποστηρίζουν την έρευνα και την καινοτομία, ε, βάση και των τοπικών ε, συνθήκων αλλά και της τοπικής οικονομίας. Γι' αυτό ακριβώ θεωρούμε ότι είναι σημαντικέ αυτέ οι πρωτοβουλίε εξειδίκευση ε, και για το αποτύπωμα του άνθρακα και για την ευφυή ε, e e, βιώσιμη μεταφορά. Όσον αφορά τώρα το κατάλογο των πόλεων, βεβαίως θα περίμενα να συμπεριληφθεί και το Μπέρμιγχαμ. Θα πρέπει σίγουρα να είναι μια εθνική διαδικασία, διότι πρέπει να υπάρχουν κριτήρια προκειμένου να αξιολογηθεί η επιλεξιμότητα της κάθε πόλης. Μία ερώτηση η οποία μου δημιουργήθηκε και αυτό ανακοινώθηκε και στην Κοπενχάγη πριν από έξι εβδομάδες από τον πρόεδρο Μπαρόζο, 5% ε, των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, θα αποτελούν αποθεματικό για τις πόλεις. Λαμβάνοντας ε, τον τρόπο με τον οποίο είναι διαστρωμένα αυτή τη στιγμή τα διορθωτικά ταμεία ε, και επειδή πολλοί θεωρούν ότι πολλοί από τη Δυτική Ευρώπη βάσει του νέου πλαισίου 2014-2020 δεν θα μπορούν να επιληθούν και τόσο πολύ από το Ταμείο Συνοχής και τα υπόλοιπα ταμεία, Ελπίζω να εξακολουθήσει να ισχύει αυτή η δέσμευση, να υπάρχει δηλαδή ένα 5% στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για τις πόλεις και να μπορούν οι κυβερνήσεις να συνεχίσουν αυτή τη διαδικασία κατάρτισης του καταλόγου των πόλεων. Και όσο πιο σύντομα γίνει, τόσο το καλύτερο, διότι ιδάλω ε, θα χάσουμε χρόνο στην ανάπτυξη του προγράμματος, κάτι το οποίο συνέβη με το προηγούμενο πρόγραμμα, ιδίω για το Ηνωμένο Βασίλειο, διότι δεν υπήρχε εφεδρικό σχέδιο και χρειάστηκαν δύο χρόνια για να εφαρμοστεί ε, και να σχεδιαστεί ένα εφεδρικό σχέδιο. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι λοιπόν ότι συμμετέχουν πλήρως οι πόλεις ε, στη ε, διαδικασία διακυβέρνησης και οι πόλεις ε, εντάσσονται στις εθνικές συζητήσεις που γίνονται για τα θέματα αυτά. Αυτό που είπε ο κύριος Βον για την ευρύτερη περιφέρεια. Εγώ μπορώ να σας μιλήσω μόνο για την περιοχή του Μπέρμιγχαμ όπου γνωρίζω τα στατιστικά στοιχεία. για περιοχές τις οποίες ε, ε, πηγαίνει κάποιος από ε, τα προάστια της εξωτερικές περιοχές στην εργασία τους εντός της πόλης. Πολλές τέτοιες δυνατότητες έχουν πολύ περισσότερη ωφέλη για την τοπική οικονομία και επειδή το Μπέρμιχαν είναι η μεγαλύτερη περιοχή στην περιφέρεια, τα ωφέλη επενδύσεων από τα διαρθρωτικά ταμεία, είτε είναι το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, είτε είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, είναι πολύ μεγαλύτερα και δεν είναι μόνο στην πόλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Πριν ε, ολοκληρώσουμε τη συνεδρίαση, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εκπροσώπους ε, των ε, περιφερειακών οργανώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, όλους εσάς φυσικά για τη συνεισφορά σας. Να σας υπενθυμίσω ότι η απογευματινή συνεδρίαση θα γίνει σε άλλη αίθουσα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή όρεξη.